Good morning everybody. Καλημέρα σας. Βλέπω ότι υπάρχει απαρτία και με χαρά κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασής μας. Όπως ξέρετε είμαστε η Περιφερειακή Επιτροπή. Έχουμε δε ως ημερήσια διάταξη αυτήν που έχετε μπροστά σας εγκρίνεται, μήπως υπάρχει κανένα σχόλιο αγαπαποίηση. Όχι, τότε εγκρίνεται. Έγκριση των πρακτικών η συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου. Ως συνήθως, αν δεν ακουστεί καμία αντίρρηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θα εγκριθούν και αυτά. Εντάξει. Στα. Δύο σύντομες ανακοινώσεις. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τη συζήτηση μετά την προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια του Στρασβούργου την περασμένη εβδομάδα. Όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι ήταν πολύ επικοδομητικά, πολύ επαγγελματικά και πολύ θετικά υπό την έποψη της πολιτικής συνοχής και των προσπαθειών μας να την καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Uh, you know that... Uh, Η πλειοψηφία που επετεύχθη κατά την ψηφοφορία ήταν εντυπωσιακή. 608 ψήφοι υπέρ. Πολύ καλή πλειοψηφία και ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες για τη στήριξή τους. Θα δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Η άλλη ανακοίνωση είναι ότι θα προσφέρω μία πρωτοχρονιάτικη δεξίωση αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασής μας στις 19 Ιανουαρίου. Για να είμαι ειλικρινής προσπάθησα να το οργανώσω για σήμερα τη δεξίωση το κοκτέιλ αλλά δεν ήταν πολύ εύκολο και γι' αυτό θα γίνει ό,τι πότε είπα. Δεν θα κάνουμε λοιπόν Χριστουγεννιάτικη γιορτή αλλά Πρωτοχρονιάτικη. Αν δέχεστε την πρόσκλησή μου βέβαια. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου. Ορίστε κύριε Βανίστελ Ρόι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα για τη δεξίωση, αλλά μήπως η γραμματεία θα μπορούσε να ελέγξει τι έγινε τελικά με το ψήφισμά μας, γιατί πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα πληροφορηθούμε από την Κομισιόν και τα λοιπά, να προσέξει δηλαδή να μας κάνει ένα χρονοδιάγραμμα. Πότε μας έρχεται η πληροφόρηση, πότε θα καθοριστεί ο χρόνος ομιλίας, τι ακριβώς γίνεται, γιατί Θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει με τις επενδύσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία. Να παρακολουθείτε λοιπόν και να μας τα πείτε γραπτός τι να αναμένουμε. Ευχαριστούμε για την πρόταση αυτή. Η γραμματεία θα προετοιμάσει αυτό το έγγραφο λοιπόν. Ήδη ετοιμάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα από την πρώτη μας συνεδρίαση τον Ιανουάριο και αναμένουμε να οργανωθεί ακρόαση της με την Προεδρία, συνεννόηση με την Προεδρία και το, την Κομισιόν των Επίτροπων. Θα το προετοιμάσουμε, θα σας τα δώσουμε όλα αυτά και αργότερα σήμερα θα σας πω για τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ της διάσκεψης των Προέδρων και των Επιτρόπων όπου έγινε μία σύντομη συζήτηση και για την πολιτική συνοχή. Θα το ετοιμα... θα Ευχαριστώ. Ξανά ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτο μας βασικό θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής με την αστική διάσταση των πολιτικών της ε και ε. Η συγγήτρια είναι η κυρία Βέστφαλ. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν πλέον σε πόλεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και κοινωνίας μας. Πολλά προγράμματα και νομοθετήματα μας αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή εκείνων που μένουν και διαβιούν στις πόλεις, αλλά συχνά δεν γίνεται αυαρκή συντονισμός. Σε ένα ψήφισμα του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις πόλεις και τον Ιούλιο η Κομισιόν ενέκρινε μια ανακοίνωση για την αστική διάσταση των πολιτικών της ε και ε. Στη δική μας έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας θα παρουσιάσουμε την ανταπόκριση του Κοινοβουλίου σε αυτή την ανακοίνωση. Σήμερα λοιπόν η εισηγήτριά μας η κυρία Βέστφαου θα μας περιγράψει τις πρώτες της σκέψεις και θα υποβάλει το σχέδιό της τον Φεβρουάριο και μάλλον θα ψηφίσουμε, θα την ψηφίσουμε την έκθεση τον Απρίλιο. Έχουμε εκπροσώπους και από την Κομισιόν, από την Γενική Διεύθυνση Περίφ, μάλιστα τον κύριο Πίσκορτς. Σας κατευχαριστώ. Κυρία Βέσφαλ, έχετε τον λόγο. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από τους ε, διερμηνείς ε, για τη φωνή μου. Παρόλα αυτά, θα ήθελα λίγο να μιλήσω για τα θέματα των ε, πόλεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε πάνω από 360 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν στις πόλεις και τα προάστια. Δύο τρίτα του ΑΕΠ παράγεται στις πόλεις. Οπότε οι πόλεις είναι κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης αλλά και ευαίσθητες στα κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα. Οπωσδήποτε τα δημογραφικά, η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι προβλήματα, τα ξέρετε. De facto, υποθέτουμε και ελπίζουμε 40-50% των ε, ποσών ε, του ΕΤΠΑ θα πάνε στις αστικές περιοχές. Εσείς είπατε, κυρία Πρόεδρε, πως ε, η σχετική συζήτηση υπάρχει ήδη εδώ και 20 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας έχει συζητήσει συχνά την θέση των πόλεων. Οπωσδήποτε το 2011 είχαμε την έκθεση Φλάζακ που ήταν πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Η ανακοίνωση της Κομισιόν για μια ατζέντα των πόλεων και οι πολλές συνεισφορές που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης κατέδειξαν πως υπάρχει η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή ατζέντα των πόλεων. Την χρειαζόμαστε γιατί πράγματι οι σωστές εξελίξεις αυτές είναι ουσιώδεις για το μέλλον μας. Το θέμα είναι τι μορφή θα έχει μια τέτοια ατζέντα, τι πρέπει να περιέχει και τι πρέπει να πετύχει. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Ο όρος πόλη πρέπει να οριστεί ε, ευρύτερα. Βεβαίως δεν ορίζει την πόλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η κάθε περιφέρεια και το κάθε κράτος ε, αναλόγως με την πολιτική του. Αυτό το οποίο δεν θέλω εγώ είναι μια πολιτική αποκλειστικά για τις μεγαλοπόλεις. Επίσης δεν θέλω αντίθεση μεταξύ αστικών και ε, αστικό περιεχόμενο και της υπαίθρου. Συχνά α, ακούγεται κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια πολιτική για τις πόλεις, δεν είναι πολιτική κατά της υπαίθρου, κατά κανέναν τρόπο. Έτσι, νομίζω πως είναι σαφές αυτό. Ακριβώς οι περιαστικές περιοχές έχουν μεγάλη σημασία για την εξέλιξη των πόλεων. Ε, εξαιρία σφύρα σας λέω, εγώ προέρχομαι από μια μεσαία πόλη 250.000 ανθρώπων στην Βαβαρία. Έχουμε θέσει εργασίας για όλους και για τις περιαστικές περιοχές. Προσφέρουμε πολιτισμό, σχολεία και περιαστική συγκοινωνία, αλλά βεβαίως είναι περιορισμένες οι αστικές περιοχές όσον αφορά, παραδείγματο χάρη, τις οικοδομήσιμες εκτάσεις. Γι' αυτό και είμαστε ευγνώμονες και εδώ πέρα θα ήθελα να αφαιρθώ στον Γιάνν Όλμπριχ το οποίος είπε πως ε, πρέπει να μιλάμε για λειτουργικές αστικές περιοχές. Αυτό ακριβώς. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό η αστική διάσταση να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αν θέλετε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα urban mainstreaming, θα έλεγα. Δηλαδή, σε όλα όσα κάνουμε, όταν διαμορφώνουμε πολιτική, να σκεφτόμαστε και τις πόλεις. Ξαναλέω, όχι ε, σε αντίθεση με την Ήπεθρο, αυτό σημαίνει πως θα έχουμε και ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Οι πόλεις, πράγματι, πρέπει αυτό το οποίο ζητάμε εδώ καιρό να έχουν περισσότερο λόγο σε αυτά που γίνονται. Πρέπει να ακούγεται καλύτερα η φωνή τους και μάλιστα ξεκάθαρα από την αρχή όχι στο τέλος της υπόθεσης. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε αυτή την αρχή της ε, Εταιρική σχέση και στα διαρθρωτικά ταμεία. Και η ατζέντα των πόλεων θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν. Τώρα το αν χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νέα νομοθεσία είναι κάτι δευτερεύον. Αλλά Εγώ θέλω να έχει ένα διαφορετικό ρόλο η, αστική πολιτική στα μυαλά και στα κεφάλια των Βρυξελών. Γι' αυτό είναι κρίμα το ότι στην επιστολή του ο Ζαν Κλοντ γιουγκερ προς την ε, νέα επίτροπο της περιφερειακής πολιτικής δεν λέει τίποτα για αστική πολιτική. Πάρα πολλά πράγματα επηρεάζουν ε, ε, όπως είπαμε, συγκοινωνίες από τη μία, προστασία του κλίματος από την άλλη. Οι πόλεις πάντα, πάντα εμπλέκονται. Μετά υπάρχει η τομεακή προσέγγιση που οδηγεί στο να έχουμε αντιφατικά μέτρα. Κάτι τέτοιο είναι θανατηφόρο για τις πόλεις. Αυτά τα βλέπουμε και στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε μέχρι πρόσφατα η ε, ομάδα που ασχολείται με τις πόλεις. Με το λεγόμενο λοιπόν urban mainstreaming θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε συνέργειες θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ομάδα δράσης εντός της Κομισιόν ε, που να ασχολείται με αυτά τα θέματα ή θα μπορούσαμε να πούμε να έχουμε έναν απεσταλμένο για τις πόλεις νομίζω πως είναι κάτι το οποίο θα έχει μέλλον έτσι ώστε κάθε απόφαση των Βρυξελών δικιά μας δηλαδή που έχει σημασία για τις ε, πόλεις να λαμβάνει υπόψη και τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Και να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρηση Πρέπει να μην επιβαρύνουμε τις πόλεις αλλά να τις αφήνουμε να διαμορφώνουν μόνες τους την πολιτική ειδικά όσον αφορά το ΕΤΠΑ, βλέπουμε πως τα κράτη-μέλη πατάνε συχνά το φρένο όταν πρόκειται να ε, διαχειριστούν μόνες τους οι πόλεις τα διαρθρωτικά ταμεία. Ενώ συχνά τα επιχειρησιακά προγράμματα εφαρμόζονται σαφώς καλύτερα στις πόλεις. Υπάρχει και το δίκτυο των ε, πόλεων στο σχετικό κανονισμό ως πλατφόρμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να τα αναπτύσσουμε αυτά και να τα δούμε, να τα συμβιβάσουμε κάπως καλύτερα. Ολοκληρώνω λοιπόν. Χρειαζόμαστε να δούμε πώς θα αναπτύξουμε καλύτερα την αστική πολιτική. Περισσότερες συνεργίες, περισσότερο urban mainstreaming μεγαλύτερη συμπερίληψη των πόλεων και σημασία στην αστική πολιτική. Έτσι χαίρομαι ιδιαίτερα για την συνεργασία και νομίζω πως με τον Γιάνν Ολμπρίχτ προσπαθήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν τα καταφέραμε όλα, αλλά νομίζω πως είμαστε σε καλό δρόμο. Χαίρομαι για την συζήτηση και με Συγχωρείτε, σπάει η φωνή μου, αλλά έχω στείλει και ένα έγγραφο που παρουσιάζω κάποιες ε, σκέψεις μου. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλά τα καταφέρατε παρά το πρόβλημα που έχετε με τη φωνή σας. Ωραία. Τώρα θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ καταρχήν τα καλά σας λόγια για την κοινή μας εργασία κατά τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να δημιουργηθεί αυτό το intergroup και να συνεχίσουμε τη συζήτηση ως προς το αστικό περιβάλλον. Σε αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, ορισμένα στοιχεία που θα πρέπει να υπάρχουν και στην τελευταία, την τελική εκδοχή του κειμένου. Να ρωτήσουμε την Επιτροπή τι πιστεύουν ως προς την αστική ατζέντα. Γίναν διαβουλεύσεις, έλαβαν γνωμοδοτήσεις και το ζήτημα είναι τι είναι αυτή η αστική ατζέντα είναι πρόταση, είναι κατευθυντήριες γραμμές ή ένα έγγραφο διαβουλεύσεων. Ποιος είναι ο τελικός στόχος της Επιτροπής. Είχαμε και το θέμα της αστικής κινητικότητας με την Γενική Διεύθυνση Τραν άρχισαν να εργάζονται επί του θέματος και μετά παρετήθηκαν τάχιστα. Ποιος είναι ο πότερος στόχος. Μην ξεχνάτε ότι η Γενική Διεύθυνση άλλαξε όνομα. Δεν έχουμε ε, Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο, αλλά και περιλαμβάνεται και ο όρος urban, δηλαδή αστικό περιβάλλον. Άρα θα δημιουργήσουμε μία αστική πολιτική, πολιτική των άστεων δηλαδή, με νέες προτεραιότητες Θα υπάρχει περιφερειακή πολιτική και υπάρχει και η πολιτική περιβαλλοντικής ανάπτυξης που άπτεται του γεωργικού τομέα. Τι θα γίνει με τις πόλεις. Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει την, θα μάλλον θα λάβει υπόψη την αστική διάσταση σε κάθε γενική διεύθυνση ή σε πολλές από αυτές. Ένα απλό παράδειγμα. Πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για τις ευφυείς πόλεις, τα ευφυή άστεα, όπου δεν συμμετέχει η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο, αλλά η Γενική Διεύθυνση των Επικοινωνιών. Αλλά ε, δυστυχώς, ενώ μιλάμε για Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο και Έρμπαν, το αστικό σκέλος εντάσσεται σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Ποιος θα είναι λοιπόν υπεύθυνο, ο τελικός υπεύθυνο θα ορίσουμε ένα πλαίσιο πολιτικής των άστεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς μπορούμε δηλαδή να υποστηρίξουμε τις πόλεις να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτή η πρόταση μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία γιατί στην Επιτροπή δεν υπάρχει ακόμα σαφής απάντηση. Η Κομισιόν έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα ως προς την αστική διάσταση με βάση το Γεωργικό Ταμείο. Χτες συμμετείχα στην συνεδρίαση για τα δημόσια μέσα μεταφορών και έγινε λόγος για ένα νέο επενδυτικό ταμείο του Γιούνκερ όπου θα υποστηριχθούν οι δημόσιες, οι αστικές μεταφορές. Ίσως η Επιτροπή κάνει πολλά για τις πόλεις χωρίς να αναφέρεται στην έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, η δική μας έκθεση θα πρέπει να αφορά ένα σαφές μήνυμα από το Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε μια σαφή διάρθρωση στην Επιτροπή για να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί και να προτείνουμε μια ευρωπαϊκή αστική πολιτική η οποία δεν θα επικεντρώνει την προσοχή στις μεγάλες πόλεις, αλλά σε πόλεις όλων των διαστάσεων και μεγεθών. Νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε κάτι το πολύ σαφές που θα διευκολύνει και την Επιτροπή. Ωραία. Ευχαριστώ. Uh, okay. Uh, Συνεχίζουμε με τους σκιώδεις. Από τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές είναι κάποιος Όχι. παρόν. Ο κύριος Ρούλ δεν είναι εδώ. Η κυρία Τόμασίτς, θα θέλατε το λόγο. Όχι, εντάξει. Okay, we, we continue. Συνεχίζουμε λοιπόν. με την κυρία Μαρτίνα Μισελς από την ΚΟΕ. Όχι, δεν είναι παρούσα. Με συγχωρείτε, ακολουθώ τον κατάλογο που έχω μπροστά μου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Βέστφαλ, γιατί παρά τα προβλήματα που έχετε με τη φωνή σας, ε, τα καταφέρνετε έτσι ώστε να εισακουστεί η φωνή μας. Και όπως είπε και ο κύριος Όλμπριχτ, θα πρέπει να έχουμε μια αστική ατζέντα, τη συζητούμε εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρειάζεται μία συνέχεια. Χρειαζόμαστε μία πιο ε, σφαιρική προσέγγιση με τη συμμετοχή των πόλεων όταν μιλάμε για νέες ευρωπαϊκές τομεακές πολιτικές, γιατί χρειάζεται η αστική διάσταση. Αυτό δεν θα οδηγήσει σε επιπρόσθετη νομοθεσία σημαίνει ότι θα αλλάξουμε την προσέγγισή μας, την ε, μέθοδο εργασίας μας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί νέες πολιτικές, νέους τρόπους διαχείρισης των ταμείων και το διακύβευμα είναι αυτό της Ευρώπης το 70-80% των πολιτών θα ζουν σε μεγάλες πόλεις μέχρι το 2050. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη, σε μια αστική πολιτική. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Βέστφαλ ότι ε, ανησυχώ κάπως, γιατί αν δούμε το όνομα της Γενικής Διεύθυνσης, αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική των άστεων. Βλέπουμε όμως ότι έχουμε έναν επίτροπο για την περιφερειακή πολιτική και στην επιστολή Juncker δεν υπάρχει καμία μνήα για τη μία πολιτική των άστεων. Μην ξεχνάτε ότι τα οικονομικά κίνητρα θα αφορούν τις ε, πόλεις του αύριο. Όταν μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη, για νέες θέσεις εργασίας, για ευημερία, χρειαζόμαστε μία ε, στιβαρή αστική προσέγγιση. Θα ήθελα η Επίτροπος, η κυρία Κρέτσου, να ασχοληθεί και με αυτή τη διάσταση, γιατί ε, έχει ξεχαστεί η πολιτική των άστεων και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλον ένα χρόνο. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία διαβουλεύσεων. Πολλοί ενδιαφερόμενοι περιμένουν την δράση της Επιτροπής. Γι' αυτό, συνάδελφοι, θα ήθελα να προβούμε σε μία σαφή δήλωση προς την Επίτροπο Κρέτσου και προς τον Πρόεδρο Γιούνκερ. Χρειαζόμαστε δράση, δεν μπορούμε να περιμένουμε για άλλον ένα χρόνο. Όταν μιλάμε για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πόλεις και της περιφέρειες για να ληφθεί υπόψη αυτή η διάσταση και να εργαστούμε έμπρακτα στις αστικές πολιτικές για τον στον τομέα της κινητικότητας, κλιματικών αλλαγών, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής διάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δεν είναι παρόσα η κυρία Μισελ, η κυρία Μάνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Βέστφαλν για τις πρώτες αυτές ιδέες. Μέχρι το Φεβρουάριο οπωσδήποτε θα γίνουν πιο συγκεκριμένες. Για εμάς τους πράσινους τα πράγματα αυτά πάνε στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής, αλλά σε μια ευρύτερη προσέγγιση για να δούμε στρατηγικά, πολιτικά και διαρθρωτικά πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το ότι οι πόλεις έχουν έναν δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με τις περιφέρειες. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε πως οι πόλεις πρέπει να εμπλέκονται νωρίς στην πολιτική διαδικασία κατά την χάραξη οδικιών, κανονισμών. Συγκεκριμένα τι άποψη έχετε εδώ πέρα. Εγώ είμαι από την Αυστρία, υπάρχει εκεί πέρα ο έλεγχος ε, της επικουρικότητας, οπότε τα περιφερειακά κοινοβούλια εμπλέκονται εγκαίρως και αν είναι μπορούν να βγάλουν μια κόκκινη κάρτα. Εμείς οι πράσινοι επίσης θα θέλαμε να δούμε κάποια στοιχεία που αναφέρατε να τα ενισχύσουμε. Αναφέρατε κάποια πράγματα, ποικιλομορφία, σύνδεση με την ύπεθρο. Δεν βλέπουμε την αηφορία, την είπατε όμως, δεν την έχετε γράψει. Πρέπει η αηφορία ακριβώς για τις πόλεις να παίξει τον ρόλο της και να ενισχυθεί και στο έγγραφο. Επίσης, η αρχή της ε, συνεταιρικής σχέσης. Ειδικά σε σχέση με το πρόγραμμα του Jean-Claude Juncker για τις επενδύσεις, ε, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε τέτοιες συνεταιρικές σχέσεις επενδύσεων και σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να συμπεριληφθεί δηλαδή ακόμη περισσότερο η κοινωνία των πολιτών ε, στην διαδικασία αυτή και Οχ, τώρα βράχνιασα κι εγώ. Να μιλήσουμε δηλαδή για community-led local programs. Εδώ πέρα έχετε κάτι πραγματάκια στην έκθεση, αλλά δεν βλέπουμε την επίδραση των νέων αυτών εργαλείων Μια ολοκληρωμένη δηλαδή αστική προσέγγιση. Πρέπει εδώ πέρα να δώσουμε λίγη ουσία τι σημαίνουν όλα αυτά. Συνολικά θετικό είναι το ότι είπατε πως το θέμα είναι ακριβώς ε, το περιθώριο ελιγμών που έχουν οι πόλεις. Όχι μόνο πολιτικά, αλλά και οικονομικά. Κοιτάξτε, εγώ είπα από τη Βιέννη μια αρκετά πλούσια πόλη, η οποία όμως ζει τα αποτελέσματα της λιτότητας και ειδικά σε ζητήματα κλίματος, κοινωνικά ζητήματα, ενσωμάτωσης, ε, γίνονται περικοπές. Και πρέπει να παραμείνει αυτή η δυνατότητα να δρούν οι πόλεις. Ε, μιλάω για ηλική ικανότητα, καθαρά έτσι. Κατά τα άλλα είμαστε ευχαριστημένοι από την εκτεσή σας, απλά θέλουμε να γίνουν κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Ντεμάτο. Καλημέρα σας. Επειδή πρόκειται για ανακοίνωση της Επιτροπής και τις πρώτες αντράσεις ε, της εισηγήτριας, θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις κοινωνικές και πολιτιστικές ε, πτυχές, δηλαδή να δούμε πώς μπορούν να αναγεννηθούν, να αναζωογονηθούν οι πόλεις. Λαμβάνοντας υπόψη και την δημοκρατική έκρηξη των πόλεων μέχρι το 2050, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το ιστορικό κέντρο πολλών ε, πόλεων και επίσης στην περιφέρεια των πόλεων που στην ουσία αποτελούν γκέτο όπου οι άνθρωποι έχουν πολύ κακή ποιότητα ζωής. Ευχαριστώ. Κύριος Λουέρ θέλει να λάβει το λόγο. Όχι, όχι. Ο κύριος Τσίκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγηση της κυρίας Βέστιχαλ και μου έκανε μεγάλη εντύπωση διότι μπόρεσε να δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το πρώτο θέμα. Το, τα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζουν σε πόλεις. Γιατί λογικά οι πόλεις θα πρέπει να κατέχουν ένα στρατηγικό ρόλο. Ένα ρόλο συντονισμού και προγραμματισμού σε σχέση με τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, τις δημογραφικές αλλαγές και αλλαγές που ανακύπτουν με βάση παλιότερα θέματα και προβλήματα και αυτή τη συγκέντρωση του πληθυσμού, κάτι το οποίο σημαίνει να, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας με μια οικονομία που δεν είναι πια σε θέση να εγγυηθεί μια θέση εργασίας και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά, υπάρχουν διαφορές ως προς τα εισοδήματα, υψηλός δείκτης ανέργειας και γι' αυτό χρειάζονται στοχοθετημένες παρεμβάσεις άμεσα. Γιατί ακριβώς αυτή η διάσταση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε τομεακό και εγκάρσιο επίπεδο. Οι πόλεις δεν μπορούν να παραμείνουν απομονωμένες σε σχέση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα πρέπει να υπάρχει η σύνδεση, μια σύνδεση των πόλεων. Εγώ προέρχομαι από τη Σαρδινία και μπορώ να πω ότι είμαστε απομονωμένοι σε εδαφικό επίπεδο. Άρα ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει η χρήση δικτύων, έτσι ώστε τουλάχιστον εικονικά να μπορέσουμε να ορίσουμε συγκεκριμένους στόχους. Όπως πολλές φορές ελέγχθη από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε το θέμα της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. θα πρέπει να λάβουμε την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διάσταση του ζητήματος. Γιατί όπως προείπα, τα δύο τρίτα του πληθυσμού ζουν σε πόλεις. και θα πρέπει να προσδώσουμε σημασία και στην αυτή διάσταση. Thank you. And the next speaker... Ευχαριστούμε. Έτεριτς. Συμφωνώ ότι οι πόλεις πρέπει να είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Μερικές λεπτομέρειες τώρα ως προς το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. με σύνδεση διαφόρων αστικών περιφερειών ώστε να γίνουν πιο ολοκληρωμένες φορολογικά και βιομηχανικά. Παραδείγματο χάρη το μείζον Βυρμίνχαμον από όπου προέρχομαι. Φύγησαν τα θέματα της αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών και μου φαίνεται ότι μια δυσκολία θα ήταν ότι αν όλα αυτά συνδυαστούν σε μία μεγάλη αστική περιφέρεια, τότε τα χρήματα των φορολογουμένων πώς θα κατανεμηθούν. Ίσως με, μέσω των τοπικών εκλογών και της θέλησης του λαού να τεθούν διαφορετικές προτεραιότητες δημογραφικά και να χαθεί. Τι η Ποιος θα κερδίσει λοιπόν η ενωσιακό νόμος ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε. Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε. Βεβαίω, η στιγμή που έρχεται μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία είναι κάτι το πολιτικό. και Βεβαίω η πολιτική στιγμή είναι ακριβώ η νέα επίτροπος. Έχουμε τώρα και 7-6 αντιπροέδρους που συντονίζουν. Οπότε το να πέφτουμε κατευθείαν στα βαθιά είναι ε, αυτό το οποίο πραγματι ήδη ε, αποφασίσαμε. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε πιο α, άμεση. Έχουμε πολλά νέα εργαλεία τώρα. Η Επιτροπή η Juncker. Πρώτα απ' όλα. Με την Τζέσικα είχαμε φοβερές ε, εμπειρίες. Και τώρα πάει στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οπότε τι γίνεται με τις πόλεις. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από δύο-τρει εβδομάδες, ε, παρουσίασαν τις προτάσεις τους τα κράτη-μέλη. 1.200 προτάσεις ε, για το σχέδιο Juncker. Πού ήταν η πόλη σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να δούμε πιο... με μια πιο κριτική ματιά τη διαδικασία όταν μιλάμε για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Τι γίνεται στην πράξη. Αν ψήσουμε, δηλαδή όταν θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση πρέπει να μας δίνει μια γενική εικόνα. Τι συμφωνήσαμε, τι κάνουμε και τι θα αλλάξουμε. Νομίζω μια καλή ευκαιρία για τις πόλεις. Συμφωνούμε πως ε, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Μπρέ, Μπρέουα, Μπρέουα σας λένε. Μπριός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα διαφωνήσω λιγάκι με αυτά που άκουσα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακατεύεται με τα πάντα και ιδίως με αυτά που δεν την αφορούν. Η εδαφική συνοχή είναι βέβαια κοινή δικαιοδοσία με τα κράτη-μέλη και αυτό δικαιολογεί τη θέση μας ως προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σας υπενθυμίζω πάντως τα εξής. Πώς μπορούμε σοβαρά να λέμε ότι θα μιλήσουμε για αστική πολιτική ενώ υπάρχουν τέτοιες ανισότητες μεταξύ πόλεων στις χώρες μέλη που είναι τρομακτικό. Μιλάτε για αστικά προγράμματα ενώ δεν είμαστε σε θέση ούτε καν μέσα σε ένα κράτος μέλος να εφαρμόσουμε μια πολιτική για τις πόλεις άξια του ονόματός της. Στη Γαλλία ας πούμε οι περιαστικές περιοχές των μεγάλων μητροπόλεων δεν τη χάνουν καμιά σημασία και κανένας μηχανισμός δεν επιτρέπει να αποκλειστεί αυτός ο αποκλεισμός. Η πολιτική αποκέντρωση έγινε αναρχικά και συνοδεύτηκε από μείωση του ρόλου του κράτους και γι' αυτό αυτές οι περιαστικές περιοχές αντιμετωπίζουν σήμερα τεράστιες δυσκολίες ως προς τη χωροταξία τους και την οικονομική τους ανάπτυξη. Είμαι δήμαρχος μιας κοινότητας 28.000 ψυχών και σας βεβαιώνω ότι δεν χρειαζόμαστε ένα ψευτοαστικό πρόγραμμα που να το έχουν επεξεργαστεί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την καθημερινή πραγματικότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία φιλόδοξη εθνική πολιτική που να ξαναδώσει πνοή στις ανάγκες, στις τοπικές ανάγκες. Άκουσα τι είπε η κυρία Βεστφάλ, μιλάει για συντονισμένη προσέγγιση για τις πόλεις. Λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι μάλλον χρειαζόμαστε μία προσέγγιση πιο δεσμευτική. Επίσης μιλάτε για συμπερίληψη των πόλεων σε όλα μας τα προγράμματα. Πάλι λυπάμαι, αλλά δεν είναι δουλειά της Ένωσης να μας επιβάλλει πράγματα, γιατί τοπικά στους Δήμους και κοινότητες υπάρχουν εκλεγμένοι εκεί άνθρωποι τοπικά που έχουν λάβει λαϊκή εντολή και αυτοί είναι οι αρμόδιοι για να εφαρμόσουν την α ή τη β πολιτική. Επίσης μας μιλάτε για νέο νόμο, μιλάτε, λέει η κυρία Βεστφάλ, το είπε. Νομίζω ότι αυτό είναι αντίθετο με την αρχή της εθνικής κυριαρχίας. Δεν μπορεί η Ένωση να παρεμβαίνει στην α ή β κοινότητα και δήμο, γιατί εμείς αρνούμαστε να μας επιβάλλουν από εδώ τέτοιου είδους προγράμματα. Αυτά είχα να σας διατυπώσω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζω την ανάγκη να προετοιμάσουμε συγκεκριμένα προγράμματα για τις πόλεις. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υπόθηκε στην προηγούμενη μας συνεδρίαση όπου έγινε μια παρουσίαση για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο για τη νέα πολιτική συνοχή 14 με 20. Και κατά την παρουσίαση τονίστηκε ότι στα λειτουργικά προγράμματα, σε στρατηγικά έγγραφα δηλαδή που γράφουν, συγγράφουν τα κράτη-μέλη, δεν λέει και πολλά για την πολιτική των πόλεων και αυτό είναι προβληματικό διότι ήταν ένα, μία από τις απαιτήσει του κανονισμού να συμπεριλαμβάνεται η αστική πολιτική σε όλα. Με κυρίο παράδειγμα την Μπολονία. Νομίζω λοιπόν ότι αφού είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι το 16 να εφαρμοστούν όλα αυτά, καλό θα ήταν να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να διευρύνουν τα στρατηγικά τους έγγραφα και στόχους ώστε να συμπεριλάβουν και την πολιτική των πόλεων. Τώρα που πρέπει να εφαρμόσουν και την αρχή της λεγόμενης smart specialization, καλό θα ήταν να προετοιμαστούν και για να συμπεριλάβουν προγράμματα για τις πόλεις, με βάση βέβαια την αρχή της εταιρικότητας, συμφωνώ για να βελτιωθούν οι προτάσεις τους και έχουμε ακόμα λίγο καιρό για να αλλάξουν τα πράγματα και να το βάλουμε και εμείς στο στρατηγικό έγγραφο. Ο στόχος δεν είναι φυσικά να καθορίσουμε εμείς να επιβάλλουμε πολιτική στις πόλεις των κρατών μελών αλλά να βοηθήσουμε τις πόλεις όχι να επιβάλλουμε να βοηθήσουμε τις πόλεις να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και αυτό φυσικά το υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ρουόλς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η δική μου άποψη επί του θέματος. Γνωρίζω τη σημασία μιας αστικής πολιτικής και ατζέντα. Όπως τονίστηκε και από την ε, εισηγήτρια και από τους ε, προλαλήσαντες, δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος ε, των κομοπόλεων και της επαρχίας. Τονίζουμε το γεγονός ότι υπάρχει ένας υπερπληθυσμός της πόλης και αυτό σημαίνει ε, απερίμωση της επαρχίας και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει ότι δηλαδή ε, οι κομοπόλεις εγκαταλείπονται. Ένας από τους βασικούς στόχους της περιφερειακής πολιτικής είναι να καταπολεμήσει τις ε, διαφορές και τις ασυμμετρίες και διατρέχουμε τον ε, κίνδυνο να τονίσουμε αυτές τις διαφορές. Βεβαίως, οι πόλεις αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. Πολλές φορές το ιστορικό κέντρο, τα ιστορικά κέντρα μετατρέπονται σε γκέτο Υπάρχει μία γκέτοποίηση των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν ο πληθυσμός να επανέλθει στα ιστορικά κέντρα των πόλεων, να μην ερημώνονται. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τύχη των μικρών πόλεων ή κομοπόλεων. Αυτή είναι μία από τις ε, βασικές μου ανησυχίες σε σχέση με την αντιμετώπιση των ασυμμετριών αυτών, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στις ε, κομοπόλεις και στα χωριά και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπρεσό. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω ορισμένες ε, παρατηρήσεις και ζητώ συγγνώμη από την εισηγήτρια γιατί δεν έφτασα εγκαίρως ε, για να ακούσω την παρέμβαση της ε, επειδή έμπλεξα στην κίνηση των Βρυξελών. Το πρώτο θέμα που φαίνεται από την ανάγνωση του εγγράφου για την πολιτική συνοχή είναι το εξή. Κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης φάνηκε ότι οι αγροτικές περιοχές ε, μπόρεσαν να αντισταθούν περισσότερο στην κρίση. Γι' αυτό και δώσαμε μεγάλη σημασία για μια πολιτική υπέρ των άστεων. γιατί τα ευεργετήματα θα πρέπει να υπάρχουν και για τα μεγάλα αστικά κέντρα που επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Επίσης, πολλοί υπενθύμησαν ότι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχουν ε, μεγάλες ε, πόλεις με μία μεγάλη περιφέρεια. Πρόκειται για τις πόλεις όπου η πολιτική των άστεων θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις περιφέρειες αυτές γιατί αυτές τις ε, περιοχές έπληξε περισσότερο η κρίση. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μπριό ότι εάν νομίζετε ότι δεν έχετε ανάγκη, τότε μπορείτε να τα καταφέρετε με δικά σας χρήματα. Αλλά νομίζω ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μεγαλοπόλων της Ευρώπης χρειάζεται μία επενδυτική πολιτική. Όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν μεγάλες ε, πόλεις που βρίσκονται πολύ κοντά σε αγροτικές περιφέρειες. γιατί σε αυτή την ε, περίπτωση τα αγορωτικά αυτά κέντρα και κομοπόλεις γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη επειδή ακριβώς βρίσκονται πολύ κοντά στα αστικά κέντρα. Δηλαδή από τη μία πλευρά μία γεωργική πολιτική θα μπορούσε να συνεισφέρει υπέρ της ε, περιφέρειας αυτής γιατί σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να κάνουμε ε, με που είναι δύσκολα διαχειρίσιμες. Αλλά στις μεγαλοπόλεις ε, γνωρίζουμε περισσότερο, γνωρίσαμε περισσότερο την οικονομική κρίση και τις ολέθριες συνέπειες της. Επίσης, τις ε, μεγαλοπόλεις θα πρέπει να τις ε, εντάξουμε στη γενικότερη περιφερειακή πολιτική. Τέλος, διαβάζοντας την ε, έκθεση περισυνοχής, θα το πω αργότερα ως σκιώδης για θέματα συνοχής, Ανακύπτει λοιπόν ότι σε όλες τις νέες μέσα σε εξαγωγικά χώρες η ανάπτυξη αφορά περισσότερο τις ε, μεγαλοπόλεις ή τις πρωτεύουσες. Ενώ τα άλλα αστικά κέντρα δεν ε, συμμετέχουν στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γι' αυτό μια αστική πολιτική δεν θα πρέπει να αρκείται στις μεγαλύτερες, πιο σημαντικές πόλεις, αλλά και στις πόλεις μεσαίου μεγέθους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ε, ανασχηματισμών, δηλαδή η βαριά βιομηχανία ε, έχει φθήνουσα πορεία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Διαφορετικά, η ανάπτυξη και οι υπηρεσίες θα περιοριστεί στις πρωτεύουσες, άρα θα εγκαταλείψουμε τα αλλαστικά κέντρα. Ιδιαίτερα ε, όσον αφορά χώρες μικρομεσαίου μεγέθους. όπου υπάρχει ένας ε, συγκεντρωτισμός της ε, υπέρ μάλλον των πρωτεγουσών. Ο κύριος Πόλτσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ την κυρία Μπράσο και τον κύριο Μπρουά και συμφωνώ με αυτά που είπαν προηγουμένως διότι <clears throat> νομίζω ότι ε, όλα αυτά μπορεί να οφείλονται και στη μετανάστευση. Ακούσαμε προβλέψεις και μπορεί να αποτελέσει η κίνηση αυτή κάτι μοιραίο για την Ήπεθρο. Όταν αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές δημιουργείται τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα για τις ε, ερημωμένες περιοχές θα ήθελα να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα της επίπτωσης των μεταναστευτικών ροών στις δημογραφικές αυτές αλλαγές. Έχουμε 6.200 κοινότητες στην Τσεχική Δημοκρατία και δεν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον δεν φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά σε μια δεκαετία μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν ριζικά και η ιδέα ότι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Τσεχία μπορεί να μετακινηθούν από την Ήπεθρο προς τις πόλεις θα ήταν κάτι καταστροφικό για τη γεωργία μας ας πούμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τέτοιου είδους αλλαγές. Φυσικά δεν θέλω να αμφισβητήσω τη σημασία που έχει ο ρόλο, τον ρόλο που παίζουν οι πόλεις αλλά πρέπει να τονίσουμε και τις επιπτώσεις που θα έχει η μετανάστευση σε αυτό. Ευχαριστώ. κυρία Βόρθ. Σας κατευχαριστώ. Εκπροσωπώ το βορειοδυτικό τμήμα της Αγγλίας όπου υπάρχουν οι τεράστιες πόλεις του Λίβερπουλ και του Μάντσεστερ αλλά και επαρχίες με μεγάλα χωριά και μεγάλο, μεγάλο ακτο, μεγάλη ακτή. Επομένως δεν μιλάω μόνο για πόλεις αλλά και για πόλεις που λειτουργούν κυρίως ως αγορές. Και δουλειά ενός ευρωβουλευτού είναι νομίζω να διασφαλίζει ότι όλα τα κέντρα του πληθυσμού είτε αραιού πληθυσμού είτε πυκνού θα ωφελούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Δικιά μας δουλειά είναι λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές αρχές, οι ηγέτες και οι επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν και αυτές, θα ωφεληθούν και αυτές από το, τη δέσμη επενδύσεων. Η Μανχεστρία και το Λίβερπουλ ε, αυξήθηκαν και αναπτύχθηκαν ακριβώς λόγω χρημάτων του Περιφερειακού Ταμείου και στην Καμβρία ε, θα ήταν απολύτως ζωτικό για τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τέτοιες επενδύσεις. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήγα και επισκέφθηκα την περιφέρεια και μας δίνουν τέτοιου είδους προγράμματα ένα, μια αναπνοή καθώς και μεγάλη περηφάνεια. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι και η δική μου εκλογική περιφέρεια και στα χωριά και στις πόλεις θα ενδιαφέρονταν πολύ τα χρήματα του Περιφερειακού Ταμείου να χρησιμοποιηθούν όπως πρέπει και θέλουν οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι τους να το διασφαλίσουν αυτό. Κυρία Κρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο γιατί η συζήτηση τώρα στο τέλος κάπου ξέφτησε. Θα γράψουμε μία έκθεση για την αστική πολιτική. Ε, δικαίως. Γιατί θέτουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Ρέγγιο, Έρμπαν και τα λοιπά προγράμματα και μια αστική πολιτική. Είναι σημαντικό αυτό. αυτό δεν σημαίνει πως παραμελούμε άλλους τομείς. Αν η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να γράψει κάτι και για την Ήπεθρο ή τη συνεργασία Ήπεθρο και πόλεων, και αυτό να το κάνουμε. Αλλά τώρα γράφουμε μία έκθεση για την αστική πολιτική και με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε. Αναμένουμε από τις πόλεις να συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή. Την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας, ε, στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Όλα αυτά είναι πράγματα που υπάρχουν, εωρούνται αν θέλετε ως ερωτήματα και περιμένουμε κάτι από την Κομισιόν. Για να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αξίζει νομίζω τον κόπο να το δούμε. και είναι πραγματικά σημαντικά αυτά τα οποία ακούστηκαν από την εισηγητρία. Τώρα τα υπόλοιπα εντάξει. Τον επόμενο χρόνο θα έχουμε μια έκθεση για τις δημογραφικές εξελίξεις γιατί είναι οπωσδήποτε ένα σημαντικό ζήτημα το ότι αδειάζουν περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι οπωσδήποτε σημαντικό. Και για την εξέλιξη της υπαίθρου και των πόλεων. Αλλά Ας μείνουμε τώρα στο θέμα μας σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Κύριο Σχέντμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αστική πολιτική έχει το εξής πρόβλημα μπορούμε να αναπτύξουμε πάρα πολύ καλά εργαλεία για την αστική πολιτική. Όλοι συμφωνούν πως πρέπει να υπάρχει μια τέτοια πολιτική, πρέπει να είναι οριζόντια και να λαμβάνει υπόψη και όλους τους υπόλοιπους ε, τομείς και να συμπεριλαμβάνεται να ενσωματωθεί στους υπόλοιπους τομείς πολιτικής. Επίσης αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Όλμπριχτ, ο λειτουργικός ορισμός οι πόλεις δεν είναι νησιά και δεν μπορούμε να τις δούμε απομονωμένες όταν μιλάμε για μια αστική πολιτική προς όφελος της ανάπτυξης τότε πρέπει και ακούστηκε αυτό να είναι σημαντική και με την ε, έξω αστική ανάπτυξη η τοπική αυτοδιοίκηση, οι διάφοροι οτά πρέπει να συνεργάζονται. Οι κάτοικοι των πόλεων πρέπει να επικοινωνούν με τις περιαστικές περιοχές. Δεν υπάρχει ένας απλός ορισμός της πόλεως ή της αστικής περιοχής Σημασία λοιπόν έχει η λειτουργικότητα. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ρεαλιστικά τις προϋποθέσεις της σωστής συνεργασίας στο τοπικό επίπεδο για να κερδίσουν και πόλεις από αυτά που πρότεινε Βρυξέλλες. Κύριε Όλμπερχ, τη ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από όσα ακούστηκαν αν μου επιτρέπετε, ε, να κάνω μια σημαντική διευκρίνηση. Η περιφερειακή πολιτική δεν είναι η πολιτική των περιφερειών, είναι η πολιτική για τις περιφέρειες. Η αστική πολιτική δεν είναι η πολιτική των πόλεων. Έτσι, γιατί κανείς δεν θέλει να α, πειράξει και να ασχοληθεί με τις πόλεις. Είναι η πολιτική για τις πόλεις. εμείς καταβάλουμε προσπάθεια για να δώσουμε κίνητρο στα κράτη-μέλη, στις κυβερνήσεις, να δώσουν περισσότερη ανεξαρτησία στις πόλεις. Αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάγκασε τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερο περιθώριο στις ε, πόλεις ε, και όχι να μπαίνουμε ξανά στα πόδια των πόλεων. Αυτό είναι κατά της επικουρικότητας. Μάλιστα. Κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Όχι. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ο κύριος Βότζισλαβ Πίσκορτς. Έχει το λόγο. Από Thank you, Madam Chair. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ μέλη της Επιτροπής σας. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τη συζήτησή σας. Αυτή τη στιγμή τελειώνουμε την σύνοψη τα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης που έχουμε κάνει από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία και συμβολές πάνω από 220 συμβολές έχουν ληφθεί και πάνω από τα μισά κράτη-μέλη μας έδωσαν τις απόψεις τους καθώς και πολλοί οργανισμοί, σύλλογοι, η Επιτροπή των Περιφερειών γνωμοδότησε, η Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή επίσης ετοιμάζει γνωμοδότηση και παραμένουμε και τη δική σας έκθεση. Επειδή ακόμα δεν τελειώσαμε την ανάλυση της δημόσιας διαβούλευσης, παρόλα αυτά μπορούμε ήδη να δούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμα χρειάζεται δουλειά για να προετοιμαστούμε καλύτερα να πράξουμε αυτά που περιμένουν από μας. Πολλοί είπαν ότι τα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να έχουν να περιέχουν αντιφάσεις και αντιφα... αρνητικές επιπτώσεις να έχουν στη ζωή των πόλεων. Μετά συζητήθηκε πώς να ληφθεί καλύτερα υπόψη, να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες των πόλεων όταν σχεδιάζεται η ενωσιακή πολιτική. Είναι όμως σωστές οι μέθοδοι μας που να μας, έτσι ώστε να μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε υπόψη της πόλης όταν κάνουμε τη στρατηγική αξιολόγηση μας. Η Επιτροπή των Περιφερειών το έχει εξετάσει αυτό σε βάθος και θα θέλαμε να γνωρίζουμε καλύτερα πώς θα μπορούσαμε πιο αποτελεσματικά να αναλύσουμε τις επιπτώσεις των προγραμμάτων μας στις πόλεις. Επίσης στη διαβούλευση φάνηκε καθαρά ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέχεια, συνοχή μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και υπηρεσιών της ε, Κομισιόν ως προς τα πόλεις. Ο κύριος Όλμπεκτ και άλλοι το είπανε. Τα παίρνουμε πολύ σοβαρά όλα αυτά υπόψη μας Έχουμε την ε, υπηρεσία για την αστική ανάπτυξη και μας δίνει αυτό τη δυνατότητα να έχουμε από πρώτο χέρι πληροφορίες, να συζητούμε για να αποφεύγουμε τις αντιφάσεις και να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια. Το όνομα της υπηρεσίας μας αστική και περιφερειακή πολιτική δεν είναι μόνο καλοπιστικό, είναι σοβαρά πράγματα. Και για να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, πληροφορούμαστε και σας πληροφορούμε και σας τακτικά για την πρόοδό μας. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι πολύ προσεκτικά θα εξετάσουμε και τη δική σας έκθεση και θα σας απαντήσουμε με σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθήσουμε αυτή την δραστηριότητα και τις προσπάθειες της Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να προετοιμάσουμε μία πολύ καλή έκθεση πρωτοβουλίας και πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση θα βοηθήσει την συζήτηση και πιστεύουμε ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα έχουμε ολοκληρώσει τις ε, διαδικασίες και κατά τους πρώτους χρόνου θα είμαστε έτοιμοι. Η κυρία Βέστφαλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η συζήτηση και οι πολλές παρεμβάσεις έδειξαν πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα ξεκάθαρα. Το είπα στην αρχή. Δεν ήταν εδώ όλοι οι συνάδελφοι. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αντιπαράθεση ε, πόλης και υπαίθρου. Μαζί πάνε αυτά, δεν είναι θέμα αντίθεσης. Δεν πρέπει να μπούμε καν σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι θέμα μεγάλου πόλεων μόνο, αφορά και τις μεσαίες και τις μικρές πόλεις και άλλα οι πόλεις είναι και κινητήρια δύναμη της κάθε περιοχής και περιφέρειας. Και ακριβώς το θέμα είναι οι πόλεις και 3.000 κατοίκους να έχουν. Ε, γιατί μπορεί να είναι πόλεις, αυτό το κρίνει όχι εμείς. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανεξαρτήτως του, ποια είναι τα μέτρα να έχουν κάποιο περιθώριο, κάποια διακριτική ευχαίρεια. Τα κράτη-μέλη λένε δεν το θέμε. Εμείς όμως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να δώσουμε αυτό το εργαλείο στις πόλεις. Αν θα το χρησιμοποιήσουν μετά είναι δικό τους θέμα, αλλά πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυτό το νόημα έχει η έκθεση αυτή. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί. Εγώ νομίζω πως θα είναι μια καλή έκθεση. Και θα έχουμε πρόοδο γενικότερα για τις πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι μία ανταλλαγή απόψεων σε μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Κάθε τρία χρόνια η Επιτροπή δημοσιεύει μία έκθεση για την πολιτική συνοχής το 2007-2013 θεωρήσαμε ότι έχει γίνει μία μείωση στο, στις δημόσιες επενδύσεις από την αρχή της κρίσης. Και αυτό τονίζει τις ανισότητες. Επίσης, ε, η πολιτική το 2014 20 θα πρέπει να σταθεί όχι στα μεγάλα έργα υποδομής, αλλά στην αποδοτικότητα της ενέργειας, τη ΜΜΕ και ούτω καθεξής. Ο κύριος Ντόιτς θα μας ε, μιλήσει για την έκθεση επιτροπής ε, και το Φεβρουάριο θα ε, μας παρουσιάσει την τελική έκθεση και θα ψηφίσουμε το Μάιο. Έχουμε εκπροσώπους από τη Γενική Ευθυνεύθυνση Ρίτζιο και Εμπλόιον, ο κύριος Άγγελ Καταλίνα Ρουβιάνες και από την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση την κυρία Κόλεβα. Άρα δίνω το λόγο στον κύριο Ντόιτς καταρχήν. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την έκθεση περί εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πέμπτη έκθεση δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποία μίλησε για τους ε, στόχους ως προς την πολιτική συνοχής μετά το 2015. Από τον Ιανουάριο του 2014 η πολιτική συνοχή της Ένωσης έχει λάβει νέα μορφή. Έχουμε τώρα ενώπιόν μας την έκτη έκθεση περί συνοχής και κατά τη γνώμη μου αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε, να δώσουμε μια νέα όθηση στην πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 75 της συνθήκης αναφέρει ότι κάθε τρία χρόνια η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει μία έκθεση στο Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και ΕΟΚΕ και Επιτροπή Περιφερειών για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην πολιτική συνοχής. Τώρα αρχίζουμε με την ανταλλαγή απόψεων ως προς την έκτη έκθεση συνοχής και τη θέση του Κοινοβουλίου ως προς την έκθεση αυτή. Η έκ εσύ ασχολείται με τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και αναλύει την πολιτική συνοχής με βάση τους στόχους της πολιτικής Ευρώπη 2020. Η πολιτική συνοχή είναι απόλυτα απαραίτητη και έχει συνεισφέρει για να ελαφρύνουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Γίνεται λόγος για την χρηματοδότηση των επενδύσεων γιατί τα κράτη-μέλη έπρεπε να προβούν σε περικοπές τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την ε, πολιτική αυτή. Χωρίς την πολιτική συνοχής η κρίση θα είχε ακόμα πιο αρνητικές επιπτώσεις. Η κρίση έχει επιβραδυνθεί ευτυχώς. Δυστυχώς όμως η ανεργία έχει αυξηθεί σε όλες τις περιφέρειες, ιδιαίτερα τις λιγότερο αναπτυγμένες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτύξουμε μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 την απασχόληση. Χρειαζόμαστε λοιπόν πραγματική πρόοδο και ανάπτυξη. Θα ήθελα να κάνω δύο βασικές ε, δηλώσεις και σε αυτό θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου. Καταρχήν, θα πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα ρευστότητας αν θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη κατά την περίοδο 2007-2013 ε, έχουμε καθυστέρηση πληρωμών 23,5 εκατομμυρίων ευρώ και αυτό βεβαίως υποσκάπτει την αξιοπιστία της πολιτικής συνοχής δεν μπορούσαμε να απαλύνουμε τις επιπτώσεις της κρίσης μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020. Η καθυστέρηση πληρωμών είναι πολύ σημαντική διότι επιβραδύνει το ρυθμό εκτέλεσης των προγραμμάτων. Ε, αυτή η καθυστέρηση πληρωμών στην περίοδο 2007-2013 οδηγεί σε καθυστέρηση ως προς την εφαρμογή των προγραμμάτων για την τρέχουσα περίοδο και φυσικά η υποβαθμίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής. Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν σημαίνει αποκλειστικά συμμόρφωση αλλά και έγκαιρη καταβολή των πληρωμών. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε και τον ρόλο της πολιτικής συνοχής. Δηλαδή συνοχή σε όλες τις περιφέρειες, ιδιαίτερα σε σχέση με τις λιγότερο αναπτυγμένες ε, περιφέρειες και αυτό σχετίζεται με την ε, τρέχουσα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές αυτό είναι ένα μέσο για να εφαρμόσουμε τους στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης 2020. Και φαίνεται ότι θα θέλαμε να βρεθούμε να λάβουμε υπόψη τους αρχικούς ε, στόχους της πολιτικής συνοχής. Έχει λοιπόν ε, σημασία να μειώσουμε τις ε, διαφορές μεταξύ περιφερειών και να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε για την ε, εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 κατά ευφυή e e και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα να μας απασχολήσει στην έκθεση είναι το εξής. Το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής είναι ύψης της σημασίας και μας ενδιαφέρει η ε, συνδεσιμότητα με το γενικότερο σχέδιο Juncker. Θα ε, ανακύψει ένα ταμείο επενδύσεων 300 δις ευρώ για να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της υποδομής και της επενδύσεις. Η πολιτική συνοχή έχει παρόμοιους στόχους. Μιλάμε για 325 δις ευρώ για την περίοδο 14-20. Γι' αυτό έχει σημασία να προωθήσουμε και το σχέδιο Juncker γενικότερα. Σε αυτό το στάδιο έχουμε τα ίδια προβλήματα διότι τα προγράμματα έχουν εγκριθεί με καθυστέρηση. Γι' αυτό η πολιτική συνοχής και η εφαρμογή της θα πρέπει να μας απασχολήσει έμπρακτα. Το 2019 θα είναι πολύ σημαντική χρονιά γιατί θα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο, μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Στρατηγική Ευρώπη 2020 και το νέο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθούν με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, την Επιτροπή Συνοχής μετά το 2020 και ούτω καθεξής. Και θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά το 2020 όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Μας ενδιαφέρει η ευημερία του ατόμου και η συλλογική ευημερία, η έκ η έκτη έκθεση συνοχής είναι πολύ συνεκτική και ασχολείται με τα αποτελέσματα, επικεντρώνεται στα αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία σχετίζονται με την υπεύθυνη διακυβέρνηση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μακροοικονομικούς παράγοντες. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια εκεί όπου υπάρχει περίπτωση αναστολής πληρωμών και πιστεύω ότι οι πολιτικοί φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κοινοβούλιο απαιτεί έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών. Η απασχόληση είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας στην έκθεσή μου και σχετίζεται και με τις ε, ΜΜΕ σε σχέση με την ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς η πολιτική συνοχή θα πρέπει να ε, διαθέτει τα μέσα για τη βελτίωση της απασχόλησης και για την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση στην ε, πολιτική συνοχής για την περίοδο 14-20 έτσι ώστε να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή χρήση των πολιτικών που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία να χρησιμοποιηθούν στην συγχρηματοδότηση και να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με ενδιαφέρει η άποψη των συναδέλφων σε σχέση με την έκτη έκθεση στην αρχή των διαβουλεύσεων και προσβλέπω στους επόμενους μήνες όπου θα συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχουν οι ε, σκιώδεις. Ε, η κυρία Μπρέσο. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια πρώτη παρατήρηση του άκουσα τον εισηγητή. Η πολιτική συνοχή έδωσε με μέχρι την κρίση για τη μείωση των διαφορών στην Ευρώπη, δηλαδή αύξηση των εισοδημάτων και μείωση των διαφορών. Το πρόβλημα είναι όμως ότι από το 2008 η κατάσταση άλλαξε άρδιν και οι διαφορές ε, μεταξύ περιφερειών ε, αυξάνονται. αυξάνονται. Και συνεπώς ε, οι στόχοι της Ευρώπης 2020 βρίσκονται πολύ μακριά από την πλήρωσή τους. Δεύτερον, μια παρατηρήση που έκανα και πριν, η κρίση έπληξε περισσότερο τις αστικές περιοχές, ενώ οι αγροτικές περιοχές μπόρεσαν να ε, αντισταθούν στην κρίση. Άρα, στα πλαίσια μιας νέας πολιτικής συνοχής θα πρέπει να ανακτήσουμε και τις δυνάμεις ως προς τις ε, αγροτικές περιοχές. Επίσης, μπορέσαμε να ανταποκριθούμε ως προς την ε, ε, σχολική παρακολούθηση, αλλά ως προς την καινοτομία επικεντρωνόμαστε στις πιο δυνατές περιφέρειες. Δυστυχώς όμως η καινοτομία δεν θα αναπτυχθεί και στις ε, πιο περιθωριακές περιφέρειες. Κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει μέσα στα πλαίσια της νέας πολιτικής συνοχής. συνοχής. Δεν θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα. Ο συνάδελφος τόνισε ότι η κρίση στα περισσότερα κράτη-μέλη υποχρέωσε τα κράτη να μειώσουν τις επενδύσεις τους και αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιφέρειες οι επενδύσεις που άπτονται της ε, πολιτικής συνοχής μειώθηκαν. Και αυτό έρχεται σε αντίφαση με μια συμπληρωματική πολιτική και όχι πολιτική υποκατάστασης, δηλαδή ναι, ναι δεν σημαίνει ότι η πολιτική συνοχής ε, δεν θα σχετίζεται με τις επενδύσεις των κρατών. Επ' αυτού του θέματος θα πρέπει να δούμε με την ε, νυν Επίτροπο πώς αυτό το θέμα θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με την νυν Επίτροπο. Επίσης η πολιτική συνοχής ναι ήταν αρχικά μια πολιτική που ασχολείται με τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, αλλά τώρα ασχολείται και με τις πλέον αναπτυγμένες περιοχές που έχουν πρόβλημα προσαρμογής προς τη νέα κατάσταση. Και αυτό αποτελεί επιτυχία και του Κοινοβουλίου, γιατί ασχοληθήκαμε για μια περιφερειακή πολιτική για όλους, ως προς το μέλλον. πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μία πραγματική εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει δεν θα σταθούμε μόνο στις περιφέρειες, αλλά όπως είπε και η κυρία Βέστφαλ και άλλοι, θα ασχοληθούμε με τις πόλεις στον προγραμματισμό της νέας πολιτικής συνοχής. υπάρχει ένας κίνδυνος ε, συγκεντρωτισμού στα μεγάλα αστικά κέντρα από τα κράτη, ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε μια περιφερειακή πολιτική και από την ε, άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. σε σχέση με τις ε, περιφέρειες που σχετίζονται με την αξιολόγηση για την εφαρμογή της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι η πρόκληση έγκυται στον ε, καλύτερο τρόπο επαλήθευσης της ε, δαπάνης των πόρων και των αποτελεσμάτων που είναι απότοκα από αυτή την πολιτική. Επίσης, η ανάπτυξη της καινοτομίας και όπως είπε και ο συνάδελφος, θα πρέπει να συνδέσουμε την πολιτική συνοχής με το πρόγραμμα Juncker γιατί το πρόγραμμα Juncker ε, επεκτείνεται σε αυτή τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης είτε στο smart grid, είτε σε σχέση με τις μεταφορές, το ευρυζωνικό σύστημα και ούτω καθεξής. Και αν όλα αυτά συνδεθούν με την ε, πολιτική συνοχή, τότε θα μειωθούν οι διαφορές στην Ευρώπη. Γιατί οι διαφορές δεν ανακύπτουν από τοπικά προβλήματα, αλλά από τις ε, δυσκολίες των πιο απομακρυσμένων και περιθωριακών ε, περιφερειών να συνδεθούν με τις κεντρικές. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί αυτή η συνδεσιμότητα με το νέο σχέδιο Juncker και την πολιτική συνοχής. Oh, and the next speaker is Mrs. Tomasic. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμασιτς. Κυρία, ευχαριστώ. Η έκθεση για τη συνοχή κάνει μια γενική παρουσίαση της προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής που είναι σημαντικός πόρος επένδυσης και ανάπτυξης στις νέες και ιδίως χώρες μέλη. Η μακρά οικονομική κρίση εμπόδισε ορισμένες περιφέρειες, πολλές περιφέρειες να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής του 2020 ενώ όπως 75% ρυθμός αναπασχόλησης για τους νέους. Το Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία είναι βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής Ευρώπης 2020 και για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία με πιο αποτελεσματικό τρόπο χρειαζόμαστε μηχανισμούς διακυβέρνησης και συντονισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που να εγγυώνται τη συνοχή μεταξύ των προγραμμάτων. την τον καθορισμό μιας νέας ομάδας εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Περίφτη της Κομισιόν που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ευκολότερα κονδύλια από προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Και ελπίζω να μπορέσουν έτσι να αντιμετωπίσουν τις καθυστερήσεις και τις, τους απαραίτητους σχετισμούς πρέπει να γίνουν μεταξύ παλαιών και καινούριων προγραμμάτων. Η Κροατία βέβαια ήρθε τελευταία και γι' αυτό καθυστερία. Ε, σε σχέση με παλαιότερες χώρες μέλη που έχουν χρησιμοποιήσει πάνω από το 50% των ε, κονδυλίων τους ενώ η Κροατία παραμένει στο 21%. Λόγω όλων αυτών όλοι οι τομείς επενδύσεων πρέπει να βασίζονται σε μια σωστά ρυθμισμένη στρατηγική που να ταυτίζει και να καθορίζει στρατηγικές προτεραιότητες και να βοηθήσει έτσι κάθε περιφέρεια να αναπτυχθεί ως το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίω, η έκθεση αυτή μας δίνει μια υποπτία της τελευταίας περίοδου, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ε, επίσης περιέχονται Έχουμε... Ζούμε μια κρίσιμη περίοδο με την ύφεση, τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων, αύξηση της ανεργίας των νέων. Αυτές είναι οι προκλήσεις Βλέπουμε λοιπόν πως οι επενδύσεις ε, πάνε από τις ε, υποδομές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην καινοτομία, νέα είδη καινοτομίας, καινοτόμα και πολιτικές κοινωνικές και ένταξης. Από την άλλη νομίζω πως εάν πραγματικά θέλουμε να θέσουμε στόχους πρέπει να τους ορίσουμε πιο συγκεκριμένα. Χρειαζόμαστε μια πιο έξυπνη προσέγγιση. Μετρήσιμη, ρεαλιστική και με χρονοδιάγραμμα. Η επόμενη λοιπόν έκθεση, η έβδομη, ελπίζω να μας δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. θα τονίσω κάποια πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, ε, αλλά αυτά θα φανούν μόνο στο τέλος. Να δούμε τι θα γίνει με τη στρατηγική, πιο συγκεκριμένα την περιφερειακή καινοτομία και την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όχι μόνο των στρατηγικών αλλά και των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν. Πρέπει να φροντίσουμε να μην είναι μεγάλο το διοικητικό βάρος και να βελτιωθεί η διαδικασία αλλά εγώ φοβάμαι όταν ακούω στην Ολλανδία πως οι διαχειριστικές αρχές ανησυχούν πως υπάρχουν πολλοί έλεγχοι και δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχουν δυνατότητες για να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να τους δώσουν λεφτά, έτσι. Οπότε, όπως όλα τα άλλα στη ζωή, το θέμα είναι να βρεθεί μια ισορροπία. και κουλίμπρε όπως λένε και στα γαλλικά. Μεταξύ ελέγχων που βεβαίως χρειάζονται, αλλά από την άλλη και να γίνεται και διαχείριση των έργων και να έχουμε ωραίες ιδέες που θα προωθήσουν την ανάπτυξη, θα μεταφραστούν σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν και τελικά θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πρέπει να τα έχουμε κατά νου αυτά. Από την άλλη δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τη συζήτηση για τη σημασία της αστικής διάστασης, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιόν να συμπεριλάβουν τις πόλεις, ε, τις αστικές περιοχές, ε, για να συμμετάσχουν στην εφαρμογή των πολιτικών. Τελευταία παρατήρηση. Έχουμε ορίσει ένα πολύ ωραίο στόχο. Ένα 5% του ΕΤΠΑ για τις πόλεις. Ένα ελάχιστο ποσό για να βοηθηθούν οι πόλεις να έχουν επενδύσεις. και βλέπουμε πως κάποιες εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την αρχή αυτή του 5% για την εμπλοκή του δημοσίου. Μα ε, όταν ορίζουμε ένα ελάχιστο ποσό, δεν σημαίνει ελάχιστο ποσό και αυτό είναι και τέλος ε, για τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές και να πούνε 5% και φτάνει Πρέπει τη στρατηγική αυτή να την έχουμε ως αφετηρία και να γνωρίζουμε πως τελικά η ε, αστική ανάπτυξη πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς γιατί και επαναλαμβάνουμε εδώ πέρα όταν μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη, ευημερία κτλ η ε, δράση αυτή βεβαίω κατά κύριο λόγο θα γίνει στις πόλεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργη σωστά το λέω το όνομά σας, ναι. Πάν σωστά, ευχαριστώ. Ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις. Η επίπτωση της κρίσης θα ήταν χειρότερη χωρίς την πολιτική συνοχή. Αυτό είναι βέβαιο. Ταυτόχρονα όμως η πολιτική συνοχή είναι από, τις Ευρωπα... τα ευρωπαϊκά προγράμματα που ε, ήταν τα πιο αποτυχημένα λόγω του χάσματος, του οικονομικού χάσματος που όλο και αυξάνεται μεταξύ κρατών. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε υπερβολικά περήφανοι για την πολιτική αυτή διότι πολλά κράτη-μέλη προετοίμασαν λάθος ή άσκημα αυτή την πολιτική συνοχή η οποία πρέπει να εφαρμόζεται από όλους αλλά όχι αποκλειστικά από το κεντρικό κράτος. Αυτή η τάση συγκεντρωτισμού ορισμένων κρατών παραγνωρίζει την περιφερειακή και κοινωνική διάσταση. Οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο και από την αρχή της διαδικασίας ώστε να μας δίνουν μια διαφορετική άποψη, την άποψή των. Η διαμεθοριακή συνεργασία ήταν από τις βασικές αξίες της πολιτικής συνοχής και κατ' μέ αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. καταστρέφεται. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ρίξουμε μεγάλη φρόνηση και προσοχή και ως προς τη σύνδεση του σχεδίου Γιούνκερ με την πολιτική συνοχής. Δεν πρέπει η σύνδεση αυτή να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό υπέρ του σχεδίου Γιούνκερ. Θέλω να επιλύσουμε το θέμα των καθυστερήσεων των ε, πληρωμών και να υπάρχει μία επικαιροποίηση όλων των στοιχείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Um, Ευχαριστώ. Ήδη ακούστηκαν πολλά πράγματα στη συζήτηση αυτή. Πρέπει στην έκθεση που κάνει το Κοινοβούλιο επί της έκθεσης να πούμε το γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα για το Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να διδαχτούμε και να δούμε πώς να είναι χρήσιμη αυτή η έκθεση στο μέλλον. Έχουμε και το πρόγραμμα του Juncker τώρα και πρέπει να διδαχτούμε από τις εμπειρίες των τελευταίων ετών. Και θεωρώ πως, όπως είπαν ήδη αρκετοί ομιλητές, η περιφερειακή πολιτική μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στην πολιτική λιτότητα των τελευταίων ετών. Κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν 90% ε, ε, των επενδύσεών τους από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Βλέπουμε λοιπόν ένα τεράστιο κενό επενδύσεων εδώ. Και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει πιο συνεκτική. Δεν είναι δυνατόν αφενός να δίνουν λεφτά και ε, από την άλλη να μην μπορούν να λειτουργήσουν κράτη, περιφέρειες και δήμοι λόγω λιτότητας. Κάποια πράγματα τώρα διαφορετικά που πρέπει να τονιστούν. Πρώτα απ' όλα η ορθή, ε, η χρηστή διοίκηση. Τα θέματα διαφθοράς ε, και τα λοιπά. Τα αναφέρει και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και είναι νομίζω ξεκάθαρο το ότι το ποσοστό σφάλματος είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να καταπολεμήσουμε την διαφορά. Μετά, σημαντικό για τους πράσινους το θέμα της πράσινης οικονομίας. Το ιδιαίτερο βάρος βεβαίως το οποίο αποδίδουμε στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν μιλάμε για αηφορία βεβαίως πρέπει να δούμε και την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοπικιλότητα. Για να μπορέσουμε να υπάρχει αυτός ο πλανήτης και για τις επόμενες γενιές. Και το επόμενο είναι η εταιρική σχέση και η εφαρμογή αυτής. Και είχαμε πάντα ακούμε διάφορα, διάφορα ειδήσει και πληροφορίες πως δεν εφαρμόζεται σωστά αυτή η αρχή. Πρέπει λοιπόν εμείς ως η αρμόδια επιτροπή να πούμε πως για εμάς η αρχή αυτή είναι βασικό κομμάτι της περιφερειακής πολιτικής. Ε, η σωστή συνεργασία δηλαδή με τους τοπικούς φορείς ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Δεν βλέπω την κυρία Ντίνολφη. Όχι, δεν είναι. Συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που προείπε η κυρία Μπρεσό και δεν θέλω να πω πολλά. Εν πάση περιπτώσει το έκτο πρόγραμμα έχει ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο. Έχει μειωθεί, έχουν μειωθεί οι δημόσιες επενδύσεις κατά 20% μεταξύ 2008 και 2013 και σε χώρες όπως η Ισπανία, Ελλάδα και η Ιρλανδία μέχρι και 60%. Γι' αυτό και η μοναδική επενδυτική πολιτική στα κράτη αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Βεβαίως η πολιτική λιτότητας υποσκάπτει την ισότητα, την εδαφική αλληλεγγύη, την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών, ιδιαίτερα στις πόλεις του Νότου. Γι' αυτό νομίζω ότι η Ευρώπη θα μας οδηγήσει στην αντιμετώπιση μιας νέας ύφεσης. Υπάρχουν λοιπόν πολύ ανησυχητικά στοιχεία γιατί με την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των δημοσίων παροχών μας οδηγούν σε μία πολιτική ύφεσης με την αμεληταία χρήση αυτών των πόρων. Τα Το πρόγραμμα Juncker είναι ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανησυχίες και επιφυλάξεις πολλών χωρών. Και θα ήθελα να πω και το εξής θα πρέπει να ε, πληρώσουμε τους καθυστερημένους λογαριασμούς. Μιλάμε για 25 δις. Άρα έχουμε καθυστερήσεις και στα λειτουργικά προγράμματα για την επόμενη περίοδο. Περιμένουμε μία αλλαγή προσανατολισμού της Ευρώπης που δεν ε, έχει ανακύψει ακόμα. Έτσι ώστε να ξαναμπούμε στο μονοπάτι της σύγκλησης. Επίσης θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο σχέδιο της ηθαγένειας. Ο κύριος ε, Σίκο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα των ΜΜΕ, διότι μετά από τις διάφορες παρεμβάσεις Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες ε, μας δίνουν τα Ταμεία Συνοχής. Και αυτό το βλέπουμε στα ταμεία συνοχής. Από 70 δις περνάμε σε 140 δις την επόμενη επταετία. Πρόκειται για πόρους προς τις ΜΜΕ κατά κύριο λόγο, διότι η οικονομική κρίση γονάτισε τις χώρες και το σύστημα παραγωγής που εκπροσωπείται από τις ΜΜΕ κατά κύριο λόγο. Χωρίς μέσα λοιπόν και χωρίς ε, διαχειριστική δυνατότητα έτσι ώστε τα προϊόντα μας να μπουν σε μια αγορά που είναι μια παγκόσμια και ανταγωνιστική αγορά. Άρα η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να σταθεί σε αυτή την ε, πτυχή. Να παρακολουθήσουμε αυτή την πολιτική συνοχής. Αυτό είναι ύψη της σημασίας γιατί τα προγράμματα είναι σημαντικά, οι πόροι επίσης, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε να τις ε, διαχειριστούμε καλά και να δούμε ποιο, ποια γλώσσα χρησιμοποιεί η Ευρώπη, διότι πολλές φορές δεν έχουμε αυτές τις κατευθυντηρίες γραμμές που συνδέουν τα διάφορα στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν μία μεγάλη οικονομική και κοινωνική ε, διαφορά και απόσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν ως προς την πραγματική πολιτική συνοχής. Και εάν όπως αναφέρει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα δούμε ποιες στρατηγικές θα αναπτύξουμε. Έχουμε καθυστερήσει. Ιδιαίτερα μην ξεχνάμε ότι η Επιτροπή αυτή είναι από κοινού νομοθέτης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται για τις πρωτοβουλίες. Δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα λειτουργικά προγράμματα και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πώς υπάρχει ανάληψη υποχρεώσεων μέσα στα πλαίσια του πολιετού σχεδίου. Νομίζω λοιπόν ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2014. Ε, θα πρέπει να μας απασχολήσουν κυρίως βέβαια οι νέοι και συμφωνώ με τον συνάδελφο ο οποίος μίλησε και προέβησε μία κριτική. Δηλαδή έχουμε πληθώρα πολιτικών αλλά μία αμεληταία πολιτική ως προς την ανεργία των νέων. Έχουμε υψηλή ανεργία των νέων κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει εδώ στην Επιτροπή μου. Thank you. And now Mr. Ο κύριος Έτεριτς τώρα. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση όπως πάντα. Θυμάμαι μια ιστορία που έλεγε ο Βάτσλαβ Κλάους για έναν Αμερικανό ακαδημαϊκό που είχε επισκεφτεί την Ευρώπη, την Τσεχοσλοβακία και ρωτούσε γιατί δεν τους αρέσει το μαρξιστικό σύστημα. Είπε υπάρχουν περισσότεροι μαρξιστές σε ένα πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας από ό,τι ως ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία. Θα μπορούσε να είχε σκεφτεί και ότι στην Ένωση υπάρχουν περισσότεροι μαρξιστές σήμερα από ό,τι στην Τσεχοσλοβακία τότε. Γιατί τι ακούμε εδώ πέρα. Όλο για ανακατανομή από τη μία πλευρά στην άλλη. Και ακούμε και επίσης για το ότι αν υπήρχε μεγαλύτερος έλεγχος από το κέντρο θα ήταν τα πράγματα καλύτερα. Αυτά μου φαίνονται γνωστά και σαν επανάληψη των λαθών του παρελθόντος και πολιτικά και οικονομικά. Φαίνεται ότι δεν παίρνουμε μαθήματα από τα λάθη μας. Φυσικά, συμφωνούμε ότι ο τρόπος εξόδου από την κρίση είναι η ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη σημαίνει μείωση του κράτους, μείωση της φορολόγησης και ελευθερία έκφρασης ώστε να μπορεί ο κόσμος να ασκήσει τη δικαιώματά του. Η δημοκρατία σε κυρίαρχο κράτος σταματάει την συνοχή που ζητάτε εσείς. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους συνοχή με κυρίαρχα δημοκρατικά κράτη γιατί έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι όλοι γι' αυτό και να το σεβόμαστε. Δηλαδή να ξέρουμε ότι η ανθρώπινη ατομικότητα μας καθορίζει όλους. Όσοι ζητάνε ενοποίηση των συστημάτων εργασίας και απασχόλησης είναι καταδικασμένοι στην αποτυχία. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για όλους, αλλά να επιτρέποντας την ατομική ελευθερία του καθενός. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε κατά της ατομικότητας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε να πω μόνο πως την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Και εκεί πέρα τονίζει πως ε, εκτός από τις επενδύσεις χρειάζονται και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να προωθηθεί η ανάπτυξη. Νομίζω πως είναι καλή αυτή η συνταγή και για την πολιτική συνοχής. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε τα χρήματά μας, τα κονδύλια μας, όχι μόνο σε επενδύσεις, αλλά και σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σε έξυπνη δημοσιονομική εξυγίανση. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με το επιχειρηματικό περιβάλλον στα κράτη-μέλη. Και άρα έχουμε συνεχή προβλήματα με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Πάρα πολύ αργή και με πολλά εμπόδια στην αγορά. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αν συγκρίνουμε τώρα το νέο σχέδιο Juncker και την πολιτική συνοχής ε, είναι δύο διαφορετικά μέσα γιατί στην πολιτική συνοχής έχουμε συγκεκριμένα ποσά και μεγάλα ποσά Βεβαίως έχουμε όλο αυτό το θέμα των ε, πληρωμών που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί, αλλά αν έχουμε 350 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό για την πολιτική σύνοχης ε, και με το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που υπάρχει στο επίπεδο των κρατών μελών, γιατί κάποιοι μίλησαν και για έναν πολλαπλασιαστή 9, έτσι λοιπόν έχουμε δυνατότητα επενδύσεων 3.000 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ. Τεράστια ποσά. Και μετά αν το συγκρίνουμε αυτό με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχουμε μόλις 5 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 8,8 δις από τον ορίζοντα 2020 ε, και το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη και τα υπόλοιπα από το περιθώριο του προϋπολογισμού. Οπότε και με τα 21 που δεν τεράστιο ποσό φτάνουμε στα 350 δισεκατομμύρια με τους ε, πολλαπλασιαστές των, πρώτων, των αρχικών 21 εκατομμυρίων. Το νέο αυτό σχέδιο λοιπόν δεν έχουμε τόσο τεράστιο δυναμικό όσο στην πολιτική συνοχής. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά η ομοιότητα είναι πως στο σχέδιο αυτό το Juncker και στην πολιτική συνοχής θεωρούμε πως για να υπάρχουν αποτελεσματικές επενδύσεις χρειάζονται πραγματικά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, που θα βασίζονται σε πολύ συγκεκριμένα έργα υποδομών. Και αυτό είπε και ο κ. Γιούνκερ και πρέπει να το συζητήσουμε ε, περισσότερο για να έχουμε πιο αποτελεσματική πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Όλμπριχτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ να υποσχεθώ στους συναδέλφους πως κοιτάξτε εμείς κάποιοι από εμάς ζούσαμε σε μαρξιστικό σύστημα σας διαβεβαιώ πως έχει μια διαφορά άμα θέλετε να σας εξηγήσω αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εκθέσεις αυτές ε, ε, και επί πέμπτης εκθέσεως προτάθηκε η νέα δομή. Υπάρχει η έκθεση προόδου που απλά αναφέρει τα αποτελέσματα και τώρα κομμάτι αυτής της έκθεσης αναφέρει τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής, ένα άλλο κομμάτι περιγράφει την νέα πολιτική. Δεν είναι λοιπόν πρόταση Απλά εξηγεί το νέο πλαίσιο της πολιτικής ε, μέχρι το 2020 και τη σχετική στρατηγική. Ενδιαφέρον λοιπόν αυτό το έγγραφο γιατί μας ε, δείχνει ποια ήταν τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών γιατί δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα υπάρχουν τα στοιχεία της νέας κατάστασης και του νέου πλαισίου, κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί υπάρχει βεβαίως ε, υπάρχουν τα έργα που έχουν μείνει πίσω, υπάρχει η νέα πρόταση Juncker και η σχέση με την συνοχή που ας το πούμε διπλωματικά είναι κάπως ενδιαφέρουσα και υπάρχουν και τα νέα αυτά στοιχεία και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος. Υπάρχει ένα λάθος εδώ πέρα στο έγγραφο της Κομισιόν. Δεν υπάρχει ελάχιστο ε, επίπεδο για τις πόλεις. Τελείως διαφορετικό το κείμενο στον κανονισμό. Δεν υπάρχει όριο ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο για τις πόλεις στον κανονισμό. Το 5% είναι απλά ε, κάτι το οποίο βρίσκεται εκεί πέρα ως υπόδειξη. Το 5% είναι ε, για τα πιλωτικά έργα, για τις ολοκληρωμένες επενδύσεις, όχι για τις πόλεις 5%. Δυστυχώς κάποια κράτη-μέλη κατάλαβαν αυτό που καταλάβατε κι εσείς, ότι θα δώσουμε 5% στις πόλεις. Και είναι τραγική η παρεξήγηση. Είναι θέμα ε, διατύπωσης ε, λοιπόν που τα κάνει πλοκά. Είναι σημαντική αυτή η παρατήρηση γιατί δυστυχώς τώρα μετά από αυτή την έκθεση πρέπει να ρωτήσουμε την Κομισιόν τι γίνεται με τα επιχειρησιακά προγράμματα, τα συμβόλαια, τα αποτελέσματα που περιγράφονται τώρα στην έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί θα ήθελα να αρκεστώ στην ιδέα ότι ο εισηγητής είπε πρόκειται μια πρώτη προσέγγιση σε αυτό το ε, θέμα που προκαλεί το ζωηρό ενδιαφέρον. Θα ήθελα να δούμε και τις ποσοστοποιήσεις το 5%, το περίφημο 5% και τη σύνδεση με το σχέδιο Juncker. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα τα βελτιώσουμε κατά τις συζητήσεις μας. Ο κύριος Ντόιτς είπε ότι ο πρώτος μου στόχος είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εύστοχο για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Και το λέω αυτό γιατί ελέγχθησαν ορισμένα πράγματα που μου δείχνουν ότι ίσως παρεκκλίνουμε από τις εργασίες μας. Κατά την ταπεινή μου γνώμη βέβαια. Άκουσα τουλάχιστον δύο φορές να γίνεται λόγος για συγκέντρωση. Δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο σύστημα επιμερισμού των αποφάσεων για περιφερειακά θέματα. Εδώ εργαζόμαστε για τους πολίτες και θέλουμε να υπάρχει συνοχή. Αυτό που θα μας απασχολήσει λοιπόν κατά την άποψή μου είναι να έχουμε μια Ευρώπη με μεγαλύτερη συνοχή μέσω της περιφερειακής πολιτικής και σε επόμενη τις συνθήκες όπως ε, υπενθύμησε ο κύριος Ντόιτς. Εάν πραγματικά το Κοινοβούλιο χρησιμοποιούσε αυτά, όλα αυτά τα δεδομένα για μία επαναφορά στο κέντρο, ένα συγκεντρωτισμό που δεν έχει καμία σχέση με την ευημερία των πολιτών, αλλά με την ε, κατανομή ε, εξουσιών, τότε δεν υπηρετούμε τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην αποτελεσματικότητα της συνοχής και να μην πούμε σε ψευδοσυζητήσεις. Thank you. Uh, yes, we'll continue. Ναι, θα συνεχίσουμε. Και σήμερα έχουμε μία πληροφοριακή συνεδρίαση με την Κομισιόν. Θα μας πει μερικά πράγματα για τη νέα πολιτική συνοχής και τις αλλαγές της. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στον κύριο Βόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον συγκητή για την έκθεσή του καθώς και γιατί δεν ξέχασε το βασικό στόχο της πολιτικής συνοχής, δηλαδή να δημιουργηθεί ισοτιμία μεταξύ των πλουσιωτέρων και πτωχοτέρων περιφερειών στην Ουαλία παραδείγματο χάρη πω που προέρχομαι υπάρχουν πολύ λίγα προγράμματα υποδομών και πολύ λίγα αναπτυξιακά προγράμματα για τις πόλεις ή προγράμματα μαθητιών που να χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Επίσης πρέπει να θυμίσω ότι Ακόμη και οι λεγόμενοι καθαροί εισφορείς ε, εποφελούνται από την πολιτική συνοχή ως αυξανόμενο, αυξημένο εμπόριο του, ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιφέρειες. Βέβαια χρειαζόμαστε τη χρηματοδότηση για να εφαρμόσουμε την πολιτική συνοχή και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα των καθυστερήσεων των πληρωμών και είναι τόσο ανησυχητικό πρέπει να μας ανησυχήσει και εμάς και τα κράτη-μέλη τα ίδια καθώς και όσους ωφελούνται διότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος καθυστερήσεων πληρωμών σημαντικών προγραμμάτων. Βέβαια, το θέμα είναι και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των σχεδίων και προγραμμάτων και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι μόνο το 10% των λειτουργικών προγραμμάτων έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα. Θα δημιουργηθούν έτσι τεράστιες καθυστερήσεις σε όλες τις χώρες μέλη και περιφέρειες και γι' αυτό νομίζω ότι ως Επιτροπή έχουμε το καθήκον να πιέσουμε την Κομισιόν αλλά και τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες ώστε τα λειτουργικά αυτά προγράμματα να εγκριθούν ως το δυνατόν πιο γρήγορα για να αρχίσει η χρηματοδότηση. Και για το μέλλον θα έπρεπε να σκεφτούμε καινούργιε διαδικασίες που να επιτρέπουν την επικύρωση των προγραμμάτων πολύ γρηγορότερα. Γιατί κάθε φορά που κατατίθενται νέα προγράμματα αρχίζουν τεράστιες καθυστερήσεις για την έγκρισή τους. Πρέπει να το δούμε αυτό στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Βαν Νίστελ και Ρόι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως έχουμε εδώ πέρα μια καλή βάση για την συζήτηση. Θα πρέπει το επόμενο 6, τους 6 μήνες να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες. Είναι μια κατάλληλη στιγμή νομίζω για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Και να τους προσφέρουμε μια νέα προοπτική. Πρέπει να διατηρήσουμε το ρυθμό που έχουμε λοιπόν και αυτό το οποίο μοιράσετε εδώ πέρα και η ομιλία είναι πάρα πολύ καλή. Κάποιες σκέψεις. Ε, βλέπουμε εδώ πέρα την συνέργεια που θέλουμε να προωθήσουμε μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Μια το, το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς μπορούν να ενισχυθούν αυτά, να ενισχύσει το ένα το άλλο. Ε, και εδώ πέρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα, την ανεργία, τις επενδύσεις ε, που πρέπει να γίνουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και από την Ευρώπη, παραδείγματος χάρη επενδύσεις προσανατολισμένες σε τομείς ανάπτυξης την ε, βιώσιμη ε, ενέργεια, την ενεργειακή μετάβαση και να έχουμε ως στόχο δημιουργία θέσεων εργασίας. Μία συμπληρωματικότητα επίσης μεταξύ ταμείων. Το οποίο πρέπει να ε, είναι πλέον ορατό στα νέα επιχειρησιακά προγράμματα. Ζήτημα το οποίο πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη, παραδείγματο χάρη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλαδή να ε, μην προσφέρουμε μόνο παρηγοριά, αν θέλετε, η προσωρινή ανακούφιση σε ένα νέο ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή δουλειά αύριο, αλλά να προωθούμε και τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Επίσης πρέπει να δούμε τη συμπληρωματικότητα με το Ταμείο της ε, Υπέθρου και τον σχετικό οργανισμό και τέλος με τα Ταμεία ε, και αυτά που αφορούν βεβαίω στη θάλασσα. Ε, ειδικά οι παράκτιες ε, περιοχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα θαλάσσια ταμεία. Αυτό θέμα να δούμε. Και βέβαια σχηματίσαμε μια νέα πολιτική έτσι. Και το είδαμε αυτό στην συζήτηση για τον ορίζοντα 2020 που είναι βεβαίω ένα ταμείο ερευνητικό, αλλά το πήγαμε προς μια κατεύθυνση υποδομών ε, και βλέπουμε πως ένα 23% ε, του περιφερειακού ταμείου πηγαίνει προς την κατεύθυνση της έρευνας και ανάπτυξης. Να δούμε λοιπόν και στην πράξη ποια είναι η δυνατότητα εφαρμογής αυτών των ε, σημαντικών πηγών χρηματοδότησης στα κράτη-μέλη. Τώρα, να έρθω λίγο στη μέσο πρόθεσμη αναθεώρηση. για την οποία τώρα ασκείται πίεση έτσι ώστε η Ευρώπη να κάνει όσα περισσότερα μπορεί να αποδώσει και η σχέση αυτή βεβαίως σημαίνει πως πρέπει και εμείς να κινητοποιηθούμε με την έκθεση αυτή. Και γεγονό είναι πως τώρα έχουμε ένα νέο σύστημα το οποίο προσανατολίζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα και έχει και τα σχετικά κριτήρια. Αν δεν εκπληρωθούν κάποια πράγματα, δεν εκταμιεύονται και τα χρήματα. Οπότε τώρα η Κομισιόν έχει έναν αντιπρόεδρο ή μία αντιπρόεδρο που, που έχει ως έργο το, την καλύτερη ρύθμιση και ε, έναν άλλον που έχει αρμοδιότητα της περιφέρειας. αλλά πρέπει πάντα να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Και βέβαια ε, το άλλο θέμα είναι ακριβώς η έλεγχη, γιατί τώρα υπάρχει αίσθηση πως ε, γίνεται έλεγχος επί των ελέγχων σε διάφορα επίπεδα και δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη από τους διάφορους εταίρους ε, στον προγραμματισμό. Δίνουμε την εντύπωση πως ε, το βασικό μας έργο εδώ πέρα είναι η έλεγχη και τελικά δεν πληρώνονται τα, τα λεφτά, κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα. και εδώ συμφωνώ με τον Τόμας Ντόιτς. Δηλαδή πρέπει να ανταποκριθούμε στις ε, υψηλές ε, προσδοκίες. Επίσης αναφέρθηκε κάπου και ο πολλαπλασιαστής. Άκουσα έναν πολλαπλασιαστή 15. Δεν ξέρω πώς ε, τα Ξέρετε αυτά τα πράγματα και πώς καταλήγεται σε αυτά. Κοιτάξτε. Θα μιλάμε για τις επιδοτήσεις, 80%-90% των επιδοτήσεων πάμε, δίνουμε τα λεφτά και περιμένουμε να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτά όμως παραμένουν επιδοτήσεις. Τι λέει τώρα το σχέδιο Juncker. Δεν έχουμε επιδοτήσεις αλλά δάνεια τα οποία πρέπει να ξεπληρώσεις. Οπότε πρέπει να επενδυθούν τα λεφτά και πρέπει να υπολογίσει κανείς ότι θα τα ξεπληρώσει κιόλας. Έτσι, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο και οπωσδήποτε διαφορετικό από τα από Είναι λοιπόν τελείως διαφορετικά τα μέσα. Ή άλλες φορές είναι εγγυήσει για έργα τα οποία εγκρίνονται και θεωρούνται σωστά. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω εγώ από την Ολλανδία είναι πως εμείς μιλάμε για ένα πολλαπλασιαστή 4 με 5, αυτό υπολογίζουμε εμείς ε, το οποίο θεωρούσαν πάρα πολύ θετικό έτσι ανά ένα ευρωπαϊκό ευρώ να έχουμε άλλα 4-5. Αλλά εντάξει, αν ε, εκεί καταλήξατε εσείς δεν έχω καμία κανένα τρολόγο να το αφισβητήσω. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο κύριος Βόλτσακ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. αυτά που είπε ο κύριος Άντρης για τον Βάτσλαβ Κλάους. Αυτά δεν τα έπαιρναν σοβαρά ούτε στη χώρα μας μετά την αμνηστία που έδωσε σε χιλιάδες εγκληματίες ως πρόεδρος. Ως προς την έκθεση του κυρίου Ντόιτς νομίζω ότι είναι πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση. για τη σύνδεση απασχόλησης με συνοχή. Αλλά επίσης θέλω να τονίσω το εξής. Το κείμενο μιλάει για τις ελλείψεις στην συμφων... στις συνεταιρικές συμφωνίες και τα λειτουργικά προγράμματα. Ερωτώ λοιπόν πώς Πώς το αποτιμά. Με ποια μέθοδο. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους υπόλοιπους. Δεν θα παρουσιάσω εδώ τα κύρια συμπεράσματα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας εδώ. Θα τονίσω όμως μόνο μερικά από τα βασικά στοιχεία που θεωρεί η Κομισιόν ζωτικά για την έκθεση αυτή. Πρώτον, πράγματι η μείωση των ανισοτήτων έχει εμποδιστεί από την κρίση και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η επίπτωση της κρίσης ήταν ασύμετρη. Γι' αυτό οι ανισότητες έχουν μεγαλώσει και φυσικά είχε ιδιαίτερες επιπτώσεις σε μερικές χώρες μέλη και περιφέρειες. Τις μετρίως ανεπτυγμένες που λέμε Οι ανισότητες όμως μειώθηκαν γενικά στις περισσότερο ανεπτυγμένες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ο λόγος για τον οποίο αυτή η ομάδα χωρών έχει πληγεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν υπήρξαν επενδύσεις εκεί. Όχι γιατί μειώθηκε η δυνατότητά τους εξαγωγών, ούτε γιατί έγινε δραστική μείωση της κατανάλωσης. Οι επενδύσεις, η έλλειψη επενδύσεων εξηγείται ασύμετρα αποτελέσματα της κρίσης. Γιατί στις χώρες αυτές έπεσαν στο μισό από ό,τι πριν από την κρίση. Και εννοώ και ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως ιδιωτικές 85% των επενδύσεων στην Ένωση είναι ιδιωτικές. Αυτό εξηγεί τα τις επιπτώσεις της κρίσης και βέβαια η πρόκληση για μας είναι πώς να επανέλθουν οι επενδύσεις που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη ιδιαίτερα για αυτές τις χώρες. Η νέα Κομισιόν τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της επαναφοράς των επενδύσεων για να υπάρξει ανάπτυξη. Μερικές ιδέες μας είναι ότι για τις ιδιωτικές επενδύσεις, όπως είπαμε και στην ανακοίνωση του Προέδρου Γιούνκερ την περασμένη εβδομάδα, υπάρχουν αποταμιεύσεις στην Ένωση που θα μπορούσαν να οθήσουν τις επενδύσεις. Το θέμα είναι όμως πώς να περάσουν από τις αποταμιεύσεις τις επενδύσεις τα χρήματα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα κίνητρα και το πλαίσιο που θα δοθεί και το πώς θα δουν οι επενδυτές τον κίνδυνο. Να μειωθεί λοιπόν η αντίληψη του κινδύνου και να αυξηθεί η κερδοφορία των επενδύσεων. Εδώ η πολιτική συνοχή έρχεται στο παιχνίδι γιατί η επένδυση σημαίνει και τη δημιουργία ως προϋπόθεση ενός σωστού οικονομικού δημοσιονομικού πλαισίου. Και αυτό θα τονίσουμε ιδιαίτερα σε καινούργια περίοδο. Συνδέοντας την πολιτική συνοχή με την οικονομική διακυβέρνηση, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κλπ. κλπ. Τονίζουμε λοιπόν ότι η πολιτική δεν αφορά μόνο τις επενδύσεις καθεαυτές αλλά και τις δημιουργίας των συνθήκων για να γίνουν επενδύσεις από τον ιδιωτικό ταμέα. Άλλο στοιχείο, οι δημόσιες επενδύσεις. Φυσικά υπήρξε μεγάλη μείωση τους και η μείωση είναι πάλι ψηλότερη στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι που το λέει και το ετήσιο έγγραφο ανάπτυξης που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν ότι η πολιτική συνοχής έχει γίνει πια η κύρια επενδυτική πολιτική αλλά μεγάλο ρόλο μπορούν να παίξουν και οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό που λέει η ετήσια αναπτυξιακή μελέτη είναι ότι μερικές φορές η δημοσιονομική πειθαρχία δεν εφαρμόστηκε όπως το είχε πει η Κομισιόν. Δηλαδή το κύριο θύμα της ήταν οι δημόσιες επενδύσεις. Αυτό πρέπει να τονιστεί, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι το η επίτευξη των στόχων της συνθήκης και της μείωσης των ανισοτήτων δεν είναι μόνο ευθύνη της Ένωσης, αλλά και των καρατών μελών και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζουν την οικονομική τους πολιτική. Το λέει η συνθήκη, το λέει, το λέει. Αυτές είναι οι κύριες ιδέες. Όσο για την απορρόφηση και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να επιταχυνθεί η, επικύρωση, η διαδικασία επικυρωση των προγραμμάτων, αλλά επίσης όχι βλάπτοντας την ποιότητά τους. Διότι ακόμη μια φορά το θέμα δεν είναι μόνο η δαπάνηση χρημάτων, αλλά με τον καλύτερο, δυνατό και αποτελεσματικότερο τρόπο για να μεγιστοποιηθεί η αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτή είναι μια από τις βασικότερες ιδέες και μαθήματα που πήραμε από την κρίση στην Ένωση και ιδιαίτερα στις λιγότερο επιτυγμένες περιφέρειές της. Αυτά είχα να σας πω αυτά. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο. Καλά. Ο κύριος Δόιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν σας ευχαριστώ μόνο λόγω φιλοφρόνησης για τη συμμετοχή σας την ενεργή συμμετοχή σας. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι μας είπε ότι έχουμε έξι μήνες να συνεργαστούμε. Ε, γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμά μας και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα θέματα στα οποία αναφέρθηκα και εκείνα τα οποία απασχόλησαν και τους συναδέλφους. Σε τρία σημεία θα ήθελα να σταθώ. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την υποστήριξή σας. Οι περισσότεροι με υποστηρίξατε τίποτα ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε σημαντικά ζητήματα που δεν είναι προσωρινά. Υποβαθμίζουν την ίδια την πολιτική συνοχή το 2014 και 2015, δηλαδή οι καθυστερήσεις πληρωμών και οι καθυστερήσεις για την αποδοχή των επιχειρησιακών σχεδίων. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις σημαντικότερες πλευρές της ε, πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να γνωρίσουμε τη συνδεσιμότητα μεταξύ πολιτικής συνοχής και σχεδίου Juncker. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να διασαφίσουμε τα πάντα που σχετίζονται με αυτό. Επίσης, συμφωνώ με τα εξής σχόλια. Η κρίση μετά το 2008 η, κρίση στην ουσία υποβάθμισε όλα τα άλλα ζητήματα, μεταξύ αυτών και την πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική. Πολλοί από εμάς βεβαίως έχουμε δεσμευτεί και ασχολούμαστε ενεργά με αυτή την πολιτική, όμως είναι γεγονός ότι η κρίση ήταν ακόμα μεγαλύτερη και ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να ορίσουμε έναν στόχο. Τα επερχόμενα χρόνια η πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Η πολιτική συνοχή δεν είναι και το μόνο μέσο... για να ανταποκριθούμε στην κρίση, να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε ορισμένα επιμέρους ζητήματα στο εγγύς μέλλον. Συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε της ΜΜΕ και να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο σε επίπεδο πολυεπίπεδης ε, διακυβέρνησης και έχει μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη ότι η έκθεση δεν είναι παρά ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Εν περιπτώσει, η έκθεση αυτή είναι αρκετά στοχοθετημένη σε σχέση με την έκτη έκθεση συνοχής. Εμείς θα ε, ορίσουμε και θα προωθήσουμε την αποδοτικότητα τη δική μας τη, ως προς την Επιτροπή Συνοχής, την πολιτική με συγχωρείτε συνοχής, μέχρι το Φεβρουάριο θα έχω δώσει τελική μορφή σε αυτή την έκθεση και ναι, ναι, ναι. θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ε, αποδοτική συζήτηση και μακρά συζήτηση και έχουμε κάποια καθυστέρηση. Έχουμε δύο επιλογές. Να αναβάλουμε το σημείο 7 για την διαδικασία απαλλαγής για σήμερα το απόγευμα μετά την ψηφοφορία ή να αναβάλουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών στο τέλος της σημερινής ημέρας. Καμία. Καμία από τις δύο επιλογές. Ωραία, συνεχίζουμε. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι μία ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης πρόσβαση των εργαζομένων στις υπηρεσίες κινητικότητας και ολοκλήρωση των αγορών εργασίας. Η Ρέγκη ε, γνωμοδοτεί και η συντάκτριά μας είναι η κυρία Νταντσίλα. η ε, ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων είναι βασική, βασικό θεμελιώδες δικαιώματα με βάση τη συνθήκη. Βασιζόμαστε στο άρθρο 46 της συνθήκης και θέλουμε να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες κινητικότητας. Η συγγήτριά μας θα μας πει ποιες είναι οι αρχικές της σκέψεις και θα παρουσιάσει το σχέδιο τον Ιανουάριο, ενώ θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο. Σωστά? Η Επιτροπή Απασχόλησης θα ψηφίσει το Μάρτιο. Έχουμε και τους προσώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μωρίν και Ακέρτς από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Κυρία Ντανσίλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε μέρα 1,1 εκατομμύρια των πολιτών τι κάνουν, ε, μεταβαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη για να εργαστούν. Επίσης, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 7 εκατομμύρια έχουν μετακινηθεί, εκ των οποίων 68% ε, είχαν μία θέση εργασίας. Αυτό γίνεται δυνατόν διότι μετακινούνται ελεύθερα και μπορούν να αναζητήσουν μία θέση εργασίας σε μία άλλη χώρα, χωρίς να χρειάζεται ειδική άδεια. Εκείνοι που διαμένουν σε ένα άλλο κράτος μέλος ε, έχουν αυξηθεί κατά 60% σε σχέση με την περίοδο 2004-2007, κάτι το αποτελεί το 3,2% του εργατικού δυναμικού η ροή της μετανάστευσης έπεσε κατά εν τρίτον λόγω κρίσης. Θεωρούμε ότι η ροή κινητικότητας μετά τη διεύρυνση οδήγησε στην αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15% κατά 1% ε, μεταξύ 2004-2009. Επίσης, σε άλλα κράτη λείπει εξειδικευμένο δυναμικό, παρόλο που υπάρχει υψηλή ανεργή. 25 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων 5 εκατομμύρια είναι νέοι. Επίσης, ε, οι θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί μέσα στα πλαίσια των επικοινωνιών, της, των τεχνολογιών και της οικολογικής οικονομίας. Γι' αυτό αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς που αναζητούν μια θέση εργασίας για να μπορέσουν να εργαστούν σε όλες ε, τις χώρες μέσα στα πλαίσια της χρήσης 25 γλωσσών μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων ε, αρμοδιοτήτων. Δηλαδή κινούνται προς επαγγέλματα όπου ε, δεν υπάρχει επαρκές εξειδικευμένο δυναμικό. Κάθε μήνα η ιστοσελίδα λαμβάνει 4 εκατομμύρια επισκέψεις και ορίζει επαφές και ένα σύνδεσμο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι νέοι. Στέλνονται 75.000 CV μηνιαίως και βρίσκονται 50.000 θέσεις εργασίας θεωρούμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε στην αύξηση του αριθμού των εταίρων μέσα στα πλαίσια του Eurvest για να ε, λάβουμε υπόψη και τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς έβρεσης εργασίας και για να πληρωθούν οι κενές θέσεις. Μέσα στα πλαίσια ενός 34% των συνολικών θέσεων εργασίας οι νέοι έχουν περισσότερες δυνατότητες μέσα στα πλαίσια της κινητικότητας γιατί εδώ λαμβάνουμε υπόψη την εργασία και τη μαθητεία, τα στάζ. Μέσα στα πλαίσια του ΕΟΡΕΣΤ εξελίσσεται η ευρωπαϊκή κοινωνία, αλλά δεν αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής ο συντονισμός και η συνεργασία μέσα στα πλαίσια του δικτύου και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Παράλληλα υπάρχουν δείγματα σε κράτη-μέλη ότι υπάρχουν ανισορροπίες στα πλαίσια των διασυνοριακών μεταφορών και κινητικότητας και γι' αυτό χρειάζονται ε, δράσεις για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους. Έτσι οι δημόσιες υπηρεσίες θα απασχολήσουν ε, το εργατικό δυναμικό και θα υπάρχει και ειδική κατάρτιση ιδιαίτερα σε σχέση με την διαβίου μάθηση πάνω από 40 ετών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και της ευφυούς επικοινωνίας. Επίσης χρειάζεται καλύτερος ε, συντονισμός για να αρθούν τα νομικά προσκόμματα για τους εργαζόμενους που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα. Γιατί πολλοί δεν δέχονται θέσεις εργασίας στην Αλαδοπή, γιατί δεν είναι καλά πληροφορημένοι και είναι ανήσυχη ως προς το, σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή την καταβολή φόρων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω λόγο στους ομιλητές. Να σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι λόγω και του χρόνου που πιέζει. Λοιπόν, κύριος Χέτσμαν. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σύντομα λοιπόν και συγκεκριμένα. Στην πρόταση του κανονισμού αναφέρεται πως η περιορισμένη κινητικότητα των εργαζομένων οφείλεται στο ότι οι προσφορές από άλλες ε, γλώσσες, ε, από άλλες χώρες δεν είναι αρκετά ικανοποιητικές ή δεν γνωρίζουν τις γλώσσες ε, οι εργαζόμενοι κτλ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή στις συνθήκες, να δούμε πώς θα συμβάσουμε καλύτερα προσφορά και ζήτηση για να καλυφθούν καλύτερα οι κενές θέσεις. Υπάρχει ένα παράδοξο στην Ευρώπη. Αφενός υπάρχει ανεργία, αφετέρου υπάρχουν κενές θέσεις που δεν μπορούν να στελεχώσουν οι εργοδότες. Πρέπει λοιπόν να συμβιβαστούν αυτά τα δύο και σε αυτό θα συνεισφέρει η καλύτερη κινητικότητα, αλλά όχι μόνο οι δημόσιοι φορείς. Όσον αφορά τώρα την περιφερειακή ανάπτυξη, το θέμα είναι και η ενισχυμένη συνεργασία καθώς και συνεργασία στις μεθοριακές περιοχές. αλλά θα μπορούσαμε να μαθαίνουμε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. στόχο έχουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες εναρμόνισης και διαμεσολάβησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόληση. Η πολιτική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρμόζεται στις προκλήσεις της ε, δημοσιονομικής ε, κρίσης. Οι ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες ε, προσελκύουν ταλέντα από όλο τον κόσμο και έτσι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των χωρών τους. Από την άλλη, η φυγή των ικανών από κάποιες άλλες χώρες επιβραδύνει την δική τους ε, ε, ανάπτυξη. Η φυγή των εγκεφάλων είναι κάτι το οποίο είναι συστηματικό. για να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις όπως η γύρανση της ομάδας εργασίας και η ανεργία ταυτόχρονα και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό της ε, κάθε χώρας και πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ε, αλλαγές στα διοδρομία των εργαζομένων, αναζήτηση καλύτερων προσόντων, καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας, ένταξη και κοινωνική προστασία με τρόπο πιο βιώσιμο. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από όλα τα κράτη-μέλη να δουν ποιες είναι οι δυνατότητες να εφαρμόσουν τις βελτιστές πρακτικές στην δική τους ε, αγορά εργασίας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε στην Ευρώπη πως τα ταλέντα μας θα μένουν στις ε, χώρες τους και θα συνεισφέρουν πραγματικά στην οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να πω κάτι εξ ονόματος της Άλντε και του κυρίου Ολιρέν. πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και να βρούμε καλύτερες δουλειές για τους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Ε, υποστηρίζω λοιπόν την ενίσχυση του δικτύου το οποίο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί πλήρως. Πολλά μπορούν να γίνουν παραδείγματος χάρη οι πληροφορίες ε, που θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ κρατών μελών και να δίδονται στα άτομα τα οποία λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ταυτόχρονα όμως να μην ε, υπάρχει περιορισμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Επίσης, ενδιαφέρουν οι συνθήκες αγοράς εργασίας από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, οπότε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα βέλτιστης χρήσης των υφιστάμενων συστημάτων. Οπότε η πρόταση αυτή πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεις και λιγότερο περιθώριο ερμηνείας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βάνα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη, έχει προχωρήσει η ώρα, εμείς υποστηρίζουμε οπωσδήποτε τη πλατφόρμα αυτή κινητικότητας ε, των ε, εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών. Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια προοπτική για τους πολίτες. Για εμάς μια σημαντική πτυχή είναι να πούμε και κάποια ξεκάθαρα πράγματα για την ε, αηφόρο απασχόληση και να προσαρμόσουμε κάπως ε, και την ε, φρασεολογία μας, να μιλήσουμε για ποιοτικέ δουλειές και τα λοιπά, όπως λέμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης, η ε, κινητικότητα δεν είναι πανάκια κατά τις ανεργίες, χρειάζεται μια άλλη στρατηγική, αλλά είναι βεβαίως ένα βασικό δικαίωμα και πρέπει να τους ε, στηρίξουμε τους εργαζομένους, αλλά δεν είναι αυτή η λύση στην ανεργία. Οι χαμηλές προσφορές επίσης ε, είναι σημαντικές. Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις προσφορές εργασίας Επίσης πρέπει να προσθέσουμε τις λέξεις μη διακριτική μεταχείριση και προσβασιμότητα ειδικά για τους αναπήρους και επίσης ε, η συμπερίληψη του τριτογενού τομέα τα ανέφερε η συγγήτρια, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμπεριληφθούν ε, όταν μιλάμε για τις δημόσιες υπηρεσίες, ε, θετικό αυτό και να συμπεριληφθούν στον τριτογενή τομέα και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ. Ο κύριος Έθριτζ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όταν κανείς έχει ορισμένες ικανότητες που δεν υπάρχουν στη χώρα του, έχει δίκιο να μπορεί να πάει αλλού για να τα ασκήσει. Είναι ζωτικό να μπορεί να μετακινείται ο εργαζόμενος. Αυτό που δεν είναι σωστό είναι να είμαστε υπερβολικά ανοιχτοί γιατί τότε έχουμε προβλήματα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που υπάρχει ανεργία των νέων ρεκόρ. Εγώ ας πούμε άρχισα να δουλεύω σε ένα ζηθοποιείο και ίσως να μην χρειαζόταν να καταφύγω σε αυτό αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω, αν ήμουν εργοδότης βέβαια, καλύτερα ειδικευμένου εργαζόμενους. Είναι ζωτικό να τα σκεφτούμε αυτά. Ο προηγούμενος μίλησε για τους καλύτερους και εξυπνότερους στους τόπους που ακριβώς χρειάζονται για να αναπτυχθεί η οικονομία. Καλύτερο αυτό να πάνε κάπου αλλού παρά να ξοδέψουν όλη τους τη ζωή ως σερβιτόροι στο Λονδίνο. Πάρα πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο αν ήξεραν τι συζητάμε θα τρόμαζαν. Ευχαριστώ. Ορίστε εσείς. Εσείς με τα γυαλιά εκεί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Γαλλία γνωρίζει πάνω από 10% ανεργία ακόμη και έχουμε πάνω από 9 εκατομμύρια πτωχούς εργαζόμενους. Μέσω της οδηγίας των αποσπασμένων δίνεται η άδεια στις γαλλικές εταιρείες να εργοδοτήσουν ξένους με συνθήκες της χώρας προέλευσης τους. Ένας Γάλλος δηλαδή που προσλαμβάνει έναν Ρουμάνο θα του δίνει μισθό Ρουμανίας και όχι Γαλλίας. Αυτό είναι σκανδαλώδες διότι συμβάλλει στον αθέμητο ανταγωνισμό μέσα στην Ένωση. Οι μισθοί λοιπόν μειώνονται και θα αυξάνεται η ανεργία για χώρες όπως η Γαλλία. Αντί όμως να αναρωτηθούμε γιατί, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει στον ίδιο δρόμο ανακοινώνοντας καινούργια τέτοια προγράμματα όπως το δίκτυο ΕΡΕΣ. Σήμερα λοιπόν Μιλάμε για ελευθερία διακίνησης μονόδρομο όμως. Για εργαζόμενους που κινούνται από την Ανατολή προς τη Δύση για να μειωθεί το κόστος εργασίας. Πρέπει να έχουμε καλύτερα και περισσότερα στατιστικά στοιχεία για την προέλευση των αιτητών ε, εργασίας. Γιατί το δίκτυο που συζητάμε διευκολύνει την πρόσληψη εργαζομένων μεν, αλλά μπορεί έτσι να δίνει και ένα αθέμητο πλεονέκτημα σε μεγάλες πολυεθνικές που προσλαμβάνουν μόνο χαμηλόμισθους και έτσι διευκολύνεται το μισθολογικό dumping μέσα στην Ένωση και για μας αυτό είναι πραγματικά σκανδαλώδες. Ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο. Επειδή πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, χωρίς το κείμενο της γνωμοδότησης, ίσως να περιμείνουμε τη γνωμοδότηση και της Επιτροπής για την επόμενη μας συνεδρία όταν θα έχουμε το σχέδιο του εγγράφου. Εντάξει, για τους εκπροσώπους της Καμισιόν μάλιστα. Κύριε Ανταντσίτα θέλετε να πείτε τίποτα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις υποδείξεις και είμαι ε, πεπισμένη ότι με την ε, τροποποίηση αυτής της έκθεσης θα έχουμε μία σωστή ένδειξη για την κινητικότητα των ε, εργαζομένων ως προς τις ανησυχίες συναδέλφων για την ελεύθερη κυκλοφορία θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή και ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις θεμελιώδεις αυτές αρχές. Επίσης, ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και να λάβουμε υπόψη την ελεύθερη κυκλοφορία και την κινητικότητα που οδήγησε στην αύξηση του μέσου ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Sorry, sorry. Um, the next... Το επόμενο θέμα είναι η απαλλαγή 2013 του Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού περιλαμβάνει την έκθεσή της για απαλλαγή της Επιτροπής ως προς την εφαρμογή του προϋπολογισμού 2013. Οι συντονιστές ε, όρισαν την Πρόεδρο για γνωμοδότηση. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Πρέπει να γνωμοδοτήσουμε πριν τις 10 Φεβρουαρίου. Σήμερα θα σας πω τι προτίθεται να κάνω. Προτείνω προθεσμία για τις τροπολογίες στις 12 το μεσημέρι, στις 11 Δεκεμβρίου, μετά μπορούμε να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο και να υποβάλουμε έγκαιρα την πρότασή, μου, την πρότασή μας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ο κύριος Αλεξάνδερ Σομόζα είναι πρόσωπος της Επιτροπής από τη Γενική Διένθυση Ρέγγιο και θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για το σχέδιο γνωμοδότησης που είναι μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες. Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής έχουμε κάνει ένα βασικό βήμα προς τα μπρος για την εφαρμογή της της πολιτικής συνοχής. Είδαμε ποιες ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες στην εκτέλεση της ε, πολιτικής και του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο τομέα. Αφού λάβαμε υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013 και την έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής επί του θέματος θα ήθελα να σας πω πώς έχει η έκθεση της Επιτροπής μας για την απαλλαγή 2013 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Επιτροπή και τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πολιτική συνοχή στο 2013 ήταν όπως τα προηγούμενα έτη. Θεωρείται από το ελεγκτικό συνέδριο ε, ως μία επιτροπή ως μια ως μια πολιτικη που οδηγεί σε σφάλματα. Το 57% των πολιτικών ε, διέπονται από σφάλματα σε σχέση με 48% τα προηγούμενα έτη. Ο δείκτης φάλματος είναι 6,9 που αποτελεί μικρή ε, αύξηση σε σχέση με το 12 που ήταν 6,8 σε σχέση με τα είδη σφάλματος που ανοιχνεύονται δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα παρελθόντα έτη. Οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων, η επιλεξιμότητα και τα δημόσια έργα είναι τομείς όπου αναγνωρίστηκαν τα περισσότερα λάθη. Το ελεγκτικό συνέδριο μίλησε για καταβολή ε, πληρωμών σε επίπεδο 37% στους τελικούς ε, δικαιούχους. Αυτό αποτελεί μια μικρή άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι πρόοδος έχει επιτελεστεί κατά την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων και να δούμε ποια είναι ε, τα ποσοστά απορρόφησης. Σε σχέση με το 12, θεωρούμε ότι η Επιτροπή ζήτησε επιπρόσθετες πληροφορίες και ως προς τις επιτόπιες οποίες έρευνες και την ανείχνευση κινδύνου βλέπουμε ότι πολλές φορές έγινε αναστολή πληρωμών. Στην ε, ετήσια έκθεση η Επιτροπή μιλά για τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέσα στα πλαίσια του ρόλου εποπτείας. Άρα το μεγαλύτερο ποσοστό ανατολής αναστολής πληρωμών, με συγχωρείτε. Και οι διορθώσεις γίνονται στα πλαίσια όπου ανοιχνεύονται σφάλματα. Από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε στους στόχους ε, της ε, συνοχής σε σχέση με την αναστολή πληρωμών θα πρέπει να γίνεται σαν ίστατο μέτρο και όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέτρα, διότι η αναστολή πληρωμών θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις ε, περιφέρειες που πλήττονται από την κρίση και για την επίτευξη των στόχων συνοχής ε, γενικότερα. Επίσης θα πρέπει να έχουμε έγκαιρη πληροφόρηση και πραγματική, πραγματικά στοιχεία και να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων έργων και της κρατικής επιδότησης. Η Επιτροπή ΡΕΓΚΙ θεωρεί ότι το 80% των δαπανών στον τομέα της διοίκησης ε, γίνονται σε επίπεδο κρατών, γίνεται σε επίπεδο κρατών. Και το ΔΕΚ θεώρησε ότι υπάρχουν σφάλματα στις συναλλαγές που θα μπορούσαν να έχουν ανιχνευθεί σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ε, οικοδόμηση μέτρων, όπως είπε και το ελεγκτικό συνέδριο, για να υπάρχει συνέπεια και αποδοτικότητα των μεθοδολογιών των κρατών μελών και βελτίωση της ε, ποιότητας και διαθεσιμότητας πληροφοριών από τις Εθνικές Αρχές στην Επιτροπή για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ενισχυμένες διαδικασίες πρόληψης, ανείχνευσης και διόρθωση φαλμάτων και παρατυπιών. Αυτά τα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή στα πλαίσια των αμοιβαίων ευθυνών, συμβαδίζοντας με την επιμερισμένη διαχείριση θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή να ορίσουν στοχοθετημένα και έγκαιρα μέτρα για να υπάρχει σωστή κατάρτιση στον τομέα του διοικητικού άχθους και να, υπάρχουν, να υπάρχει προσωπικό με δεξιότητες. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να μας μιλήσει για τα αυτά αποτελέσματα μετά από την αρμοδιότητα των ε, φορέων σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές. Αυτά εντάχει της γνωμοδότησης που έχετε ήδη στα χέρια σας. Είμαι ε, το όριο των λέξεων στο σχέδιο γνωμοδότησης δεν μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε πολλές προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα σχόλιά σας και τις ε, τροπολογίες σας. Κύριε Όλμπερχτ, έχετε το λόγο. Δεν το ζήτησα, αλλά είναι σκιώδης Μία σύντομη παρατήρηση. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο πώ εκφράζονται οι διάφορες επιτροπές. Η Επιτροπή Πολιτισμού πάντα λέει δυστυχώς κτλ. τα η δικιά μας Επιτροπή είναι παραδοσιακά θετική για τα λάθη. Λέμε πως δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα, αλλά να βρούμε κάποια καλά σημάδια στην πολιτική συνοχή, λέγοντας πως η κατάσταση δεν χειροτέρεψε το επίπεδο σφαλμάτων τα τελευταία χρόνια πέφτει. Τότε θα πρότεινα να δοθεί ο δικός μας ο χαρακτήρας της Επιτροπής μας. Αυτά, δεν έχω κάποιο σχόλιο για όσον αφορά την ουσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μόνος. Ευχαριστώ. Επίκαιρο το θέμα διότι τη Δευτέρα θα προεδρεύσω μια συνεδρίαση σε Επιτροπή Ελέγχου του Προεπλογισμού με τον Αρμόδιο Επίτροπο. Και πράγματι, αν σε διαφορετικό κλίμα θα γίνει η συζήτηση, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αποτελείται από ανθρώπους που πάντοτε θέτουν προβλήματα και βρίσκουν προβλήματα να συζητήσουν. Όσο για την γνωμοδότησή σας, Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα ήθελα να κάνω και μερικά πρόσθετα σχόλια. Ένα είναι να τονίσω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ λαθών και απατών. Εμείς μιλάμε για λάθη και όχι για απάτες. Όπως για την πολιτική των προμηθειών, για τα διοικητικά, όπως ότι δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο σωστά κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για λάθη και όχι για απάτες. Η απάτη αφορά λιγότερο από 2% στον προϋπολογισμό και πολλά κράτη-μέλη θα ήθελαν να έχουν τόσο χαμηλό ποσοστό. Φυσικά θέλουμε να μειωθεί και το ποσοστό αυτό και το ποσοστό των λαθών. Κάθε χρόνο βρίσκουμε ότι πολλά από τα λάθη οφείλονται στα συστήματα και τις διαδικασίες και τον πολύπλοκο χαρακτήρα τους για τον οποίο παραπονούνται πολλές φορές οι ωφελούμενοι. Επίσης νομίζω πρέπει να τονίσουμε όσο μπορούμε το ρόλο των χωρών μελών. Οι χώρες μέλη είναι υπεύθυνε για 80% της δαπάνησης των κονδυλίων και τα περισσότερα από αυτά τα λάθη θα έπρεπε να είχαν ταυτιστεί και διορθωθεί από τα ίδια τα κράτη-μέλη πριν από την Κομισιόν. Να χρησιμοποιηθεί λοιπόν αυτή η δυνατότητα των χωρών μελών. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ταυτίσουμε ποια είναι τα κοινά προβλήματα, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να τα διορθώσουν, ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη που έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Κάθε φορά 5-6 κράτη-μέλη είναι πάντοτε τα ίδια υπεύθυνα για τα περισσότερα λάθη, να τα βοηθήσουμε τα κράτη αυτά. Με, τη, με διοικητικό τρόπο να τους δώσουμε παραδείγματα βελτίστων πρακτικών από αλλού και να τους βοηθήσουμε με το δημοσιονομικό τους έλεγχο που πολλές φορές είναι προβληματικά. Μιλάω πάντα για τα κράτη που πράττουν τα λάθη και πρέπει και να τα διορθώσουν. Τέλος, η αποτελεσματικότητα. Μιλάμε για το αν δαπανούνται σωστά τα χρήματα, αλλά πρέπει να δούμε και αν ε, δαπανούνται αποτελεσματικά. Να διασφαλίσουμε ότι ναι μεν σωστά δαπανούνται, αλλά και αποτελεσματικά. για όφελος ολόκληρων περιοχών και περιφερειών και όχι μεμονωμένων πολιτών. Θα κάνω μερικές τροπολογίες στην δρομοδότηση, όχι πολλές, γιατί γενικά συμφωνούμε με το περιεχόμενό της. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μιλάω από τον κύριο Νίκολσον, κύριε Λιάρα. Σύντομα. Να συμφωνήσουμε με κάποια σχόλια του Ντέρεκ ειδικά για το πώς θα κοιτάξουμε την απόδοση. Αυτό είναι πολύ πολύτιμο και είναι κάπως αιτία απογοήτευσης όταν θεωρούμε ότι εξοδεύτηκαν σωστά τα χρήματα και εννοούμε βασικά ότι συμπληρώσαμε σωστά τα έντυπα, όχι ότι είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς θεωρούμε πως πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ του να εργαζόμαστε αποτελεσματικά εντών των διαδικασιών αλλά και μια ευρύτερη συζήτηση για αυτούς τους προϋπολογισμούς και ειδικά για τις μεταφορές από χώρε που είναι καθαρής φορής δηλαδή δίνουν τα λεφτά τους, επιστρέφονται και μετά δίνουν και λογαριασμό και δεν μου φαίνεται λογική χρήση των δημοσίων κονδυλίων αλλά και εντός των στενότερων πλαισίων που είχαμε στο παρελθόν. Συμφωνώ με κάποια πράγματα που είπε ο Ντέρεκ και σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Είναι δύσκολο το όνομά μου να το προφέρει κανείς. Ε, θα μιλήσω κρατικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας ε, να τονίσω πως ε, η διαφάνεια στην χρήση των κονδυλίων πρέπει να είναι βασική αρχή που θα μας καθοδηγεί. Η πολιτική συνοχή συχνά υφίσταται κριτική και ακούμε πως ε, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χρήσης των κοντιλίων γιατί επηρεάζει την ίδια την πολιτική συνοχή. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την διοικητική ικανότητα των χρηστών και μετά βεβαίως πρέπει να δούμε πώς επηρεάζεται έτσι η ποιότητα ζωής στις πόλεις. Υπάρχουν διάφοροι νόμοι περί δημοσίων προμηθειών και μετά δεν συμβάζονται με αυτά εθνικές δηλώσεις. Έχουμε λοιπόν κάποια καλά αποτελέσματα από τις εθνικές δηλώσεις, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα οικονομικά μας. Συχνά τα κράτη-μέλη βλέπουν κάποιες ελλείψεις στην νομοθεσία τους και συχνά υπάρχουν κάποιες ερμηνείες ε, ε, που δημιουργούν ε, ζητήματα κακοδιαχείρισης. Συχνά οι διαγωνισμοί και οι προκηρύξεις τους δεν ταιριάζουν ακριβώς με αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά υπάρχουν και κρατικές επιδοτήσεις. Θα θέλαμε λοιπόν η Κομισιό να κάνει καλύτερους επιτόπιους ελέγχους για να έχουμε καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Θεωρώ πως εμείς ως Επιτροπή πρέπει να ζητήσουμε ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των κρατών μελών, ειδικά όσον αφορά τις δημόσιες προκήρυξεις και έτσι θα υπάρξει μείωση των σφαλμάτων και της απάτης και πιο αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων, κάτι που μας συμφέρει όλους. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίξατε το έργο μας επί της γνωμοδότησης αυτής. Οι εμπειρίες αυτές ήταν επικοδομητικές και νομίζω πως οι προθεσμία και τροπολογίες είναι το μεσημέρι της 11ης Δεκεμβρίου. Ωραία. Οπότε τελείωσε το πρώτο τμήμα της συζήτησής μας και θα ζητήσω από τους συντονιστές να παραμείνουν για τις συνεδρίες των συντονιστών. Thank you. See you later.